All right, dear colleagues, uh, I would suggest that we start, that we... Ο Πρόεδρος, συνάδελφε, να αρχίσουμε, να δούμε την ημερησία διάταξη της σημερινής μας συνεδρίασης. And I welcome you. Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή δημοσία συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρόκειται περί ακροάσεως Πρώτα-πρώτα, θερμά καλωσορίσματα στον ε, Επίτροπο κύριο Λεβαντόφσκι, τον Επίτροπο τον Αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε και θα πρέπει να δούμε Καλώς ήρθατε και οι προσκεκλημένοι μας, τα μέλη του πάνελ, οι καθηγητές και το, θέμα στο οποίο θα στην προσοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο για την Επιτροπή μας, αλλά είναι σημαντικό για όλα τα όργανα. οπότε η στρατηγική που ξεκίνησε το 2000, ε, αναδομήθηκε το 2005, εξελίχθηκε στην στρατηγική ενώ το 2020 το 2010. Κάτι το οποίο είναι το βασικό ε, πόνημα της Επιτροπής του κ. Μπαρόσο. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος το να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, ε, η οποία να είναι βιώσιμη, να καλύτερη απασχόληση, να βασίζεται στη γνώση και όλοι γνωρίζουμε ότι η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 έχει ε, ακυρώσει κάποια θετικά αποτελέσματα του 2007 και του 2008. Οπότε δεν χρειάζεται να να το εξηγήσουμε τώρα, ότι αυτό το όραμα αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Οπότε και η σημερινή ακρόαση είναι κάτι το οποίο έρχεται στην ώρα του. Διότι μπορούμε τώρα λίγο πριν τις εκλογές να κάνουμε έναν απολογισμό. Η στατική αυτή πέτυχε. Η πολιτική μας αποτελεί μια προσθεμένη αξία στις πολιτικές των κρατών μελών. ή σημειώθηκε σύγκληση των οικονομιών. Και πρόκειται για κάποια ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να θέσουμε. Και αυτό έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των ε, πολιτικών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής ε, ακρόασης και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν οι προσκεκλημένες να δώσουν τις απαντήσεις. Βεβαίως, ε, τονίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Επιτροπή μας ως θέμα. Θα δούμε επίσης, αυτό είναι ο ρόλος μας, πώς έχουν αναλωθεί τα χρήματα των φορολογουμένων. Γι' αυτό να το εξετάσουμε με την διαδικασία της απαλλαγής πολύ προσεκτικά. Σύμφωνα με τη συνθήκη, ε, έχουμε να κάνουμε με την διαδικασία συμμόρφωσης όσον αφορά την νομιμότητα, κανονικότητα, και το επίπεδο σφαλμάτων και επίσης την δήλωση DAS και την ε, προσέγγιση των επιδόσεων ε, εκτέλεση του προπολογισμού. Οπότε και εμείς είπαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδώσει αυτού του είδους την αντίληψη, το πνεύμα των επιδόσεων για να μπορούμε να κάνουμε την αξιολόγηση βάσει του άρθρου 318, Το ώστε αυτή η αξιολόγηση να συσχετιστεί με του βασικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και εμεί ρητά έχουμε παραπέμψει στου στόχου τη στρατηγική του 2020. Εκείνη η έκθεση Γκάιερ όσον αφορά την ε, παραγωγή του 2011 και η προσωπική μου έκθεση όσον αφορά τι επιδόσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή του προπολογισμού χρειάζεται μια καθαρή έποψη των στόχων επιτευγμάτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε τις εξελίσεις και να χαράσουμε τις πολιτικές εγκαίρες. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει με σοβαρότητα ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί και να μπορέσει να έχει μια βιώσιμη ε, ανάπτυξη που δεν περιθωριοποιεί κανένα. Θεωρώ ότι αυτά έλαβε υπόψη η Επιτροπή γιατί το σχέδιο προηγούμενου του 2014 το 50,7% είναι κονδύλιο που συνδυάζει με την πολιτική ενόψη του 2020. Πάντως θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να συνοδευτεί από μια ανάλογη εξέλιξη στην διαμόρφωση του προπολογισμού. Είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας να συμμετάσχουν τα θεσμικά όργανα και το Ελληνικό Συνέδριο, ούτω ώστε να μπορούμε να δούμε πώ θα καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα δράση. Αυτό θα διευκολύνει την αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επίση την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μακρόπνο έργο και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιδράσει θετικά στις απόψει του Κοινοβουλίου. Στα όσα είπαμε τον Ιούλιο του 2013 και επαναδιατυπώσαμε σε πολλές ε, περιπτώσεις. Έκτοτε, μια που δεν έχουμε έναν προϋπολογισμό που να βασίζεται στις επιδόσεις, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να μην λαμβάνει υπόψη το τι πετύχαμε στο παρελθόν, με ποια μέσα πολιτικής, ποια εργαλεία, με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε στη θέση μας να πράξουμε έτσι σήμερα. Επομένω, θα πρέπει να συζητήσουμε την στρατηγική τη Λισαβόνα και με χαρά, με αυτή την εισαγωγική παρατήρηση, θα δώσω το λόγο στην συγκεντριά μας, την κυρία Γκρέσλερ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους ομιλητές και πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν εύκολο να λάβουμε τη δέσμευσή σας ότι θα έρθετε, διότι ο τίτλος της ακρόασης, η στρατηγική της ε, Λισαβόνας, ε, για πολλούς ε, πια δεν σημαίνει τίποτα. Πιστεύω όμως ότι στα 17 χρόνια που εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική από το 2002, το 2010 βέβαια επιλέχθηκε η μετεξέλιξη και αυτής της ε, στρατηγικής ε, ε, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου διατέθηκαν 1,5 δις ευρώ στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής και το ερώτημα είναι τι λάβαμε ανταυτού. Το αποτέλεσμα θεωρούμε ότι είναι ότι υπάρχει ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερη κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει να περάσουμε σε μια κοινωνία η οποία θα βασίζεται στη γνώση. Αυτό είναι ένας από τους τρεις πυλώνες. Ο δεύτερος είναι ο εξυγχρονισμός του κοινωνικού μοντέλου και ο τρίτος πυλώνας είναι η αηφόρος ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ το τι ακριβώς έγινε από όλα αυτά τη στιγμή που είχαν τεθεί και συγκεκριμένοι στόχοι. Πρόκειται λοιπόν για μια ακρόαση η οποία έχει ως στόχο να δείξει τι ακριβώς επιτύχαμε με τη στρατηγική της Λισαβόνας, τι μάθαμε και πώς ακριβώς πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 έτσι ώστε τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά από ό,τι μέχρι τώρα. Ορισμένα κράτη, οι βόρειες χώρες, ε, η Ολλανδία και η Ευστρία τα πάνε καλύτερα, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η δική μου η χώρα και αυτές μια χαρά τα πήγαν, άλλες πάλι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν περισσότερα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διερωτηθούμε τι επιτύχαμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε με μια τέτοια στρατηγική. Γι' αυτό λοιπόν ε, τα ερωτήματα που θέτω είναι κατά πόσον ε, μπορούν διαφορετικά κράτη να επιτύχουν μια ενιαία δομή. Υπάρχει βέβαια και η μέθοδος ε, του ανοιχτού συντονισμού που ήταν ένα από τα δύνατα σημεία της πολιτικής της Λισαβόνας. Τι πρέπει να μάθουμε έτσι ώστε η Ευρώπη 2020 να είναι πραγματικά επιτυχημένη. Κατόπιν, όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε οι στόχοι αυτοί να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο από ότι μέχρι τώρα. Δηλαδή, αντί να χρηματοδοτούμε περί τι πολυτέλεια, τι ακριβώς μπορεί να προκύψει από την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει η χρήση των κονδυλίων να βρίσκεται, να είναι συμβατή με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, ποιος θα έχει τελικά την γενική επισκόπηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και όλα αυτά τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Πρέπει να διερωτηθούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αντί να περιμένουμε λοιπόν να υποβληθούν νέες προτάσεις, καλύτερα να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει με τις παλιές. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια για αυτή σας την εισαγωγή και θέλω να πω ότι όσοι διαρωτώνται τι ακριβώς έχει γίνει με τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα και οι πιο δημοφιλοί στην πολιτική. Καλώς όρισα ο Ζώμης των Τεφρένη που προέρχεται από το Ίδρυμα Σεν Λουί των Βρυξελών. Καλώς ορίζει και στα γερμανικά. Εκτός μικροφόνου. Oui, je vais donc euh, essayer de structurer. Euh... Για να δούμε πρώτα πρώτα το πλαίσιο στο οποίο έχω προετοιμάσει την ομιλία για, ε, ε, φυσικά σε σχέση με το πώς και αυτή η συνήθεια της αγώνας. Οπότε πρώτα πρώτα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το one size fits all. Δηλαδή θέλουμε το, να δούμε το, ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί υπόψη η ετερογένεια στις οικονομίες των κρατών μελών. Στη συνέχεια θέλω να δούμε μια άλλη ανάλυση της σημερινής καταστάσεως ιδίω ε, κατόπιν ε, του 2009 που ξεκίνησε η κρίση. Να σας πω τι γίνεται με την Ευρώπη 2020, ε, μετά δηλαδή την συνδίκη της Λισαβόνας, κάτι το οποίο δεν έφερε διόρθωση στην πορεία μας, γιατί είχαμε διαφορετικές διαδρομές της οικονομίας. Άλλα γίνανε στην Βόρεια Ευρώπη και άλλα γίνανε στην περιφέρεια. Έχουμε βέβαια και κάποιες χώρες της περιφόρειας που εξαιρούνται και έχουν καλές επιδόσεις και οπότε να δούμε σε ποιο πλαίσιο διαμορφώθηκε η στρατηγική της Λισαβόνα. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90 η Ευρωπαϊκή Στρατηγική εστόχευε στο να βελτιώσει την οικονομική ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς γιατί οπότε είχαμε αυτή την ανάλυση που είχε γίνει εδώ και δεκαετίες ε, και είχαμε επομένω τις πολυεθνικές, τις αμερικανικές οι οποίες ως πλεονέκτημα είχαν το ότι μπορούσαν να δράσουν στην εσωτερική τους αγορά, να κάνουν οικονομίες κλίμακος, όμως από την άλλη μεριά ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ήταν κατετιμημένος με τους ε, δασμούς και με διάφορους ε, ε, άλλους φραγμούς που δεν μπορούσαμε να πετύχουμε λόγω αυτών της οικονομίας κλίμακος. Οπότε κάναμε την ενιαία αγορά και από το 1968 καταργήθηκαν οι δασμολογικοί φραγμοί και οι τεχνικοί φραγμοί, οι τεχνολογικοί ε, έχουμε όμως εδώ πέρα πάρα πολλές μικρές ε, μονάδες που παράγουν αντίθετα με την Αμερική οπότε εμείς δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις οικονομίες κλίμακος οπότε έχουμε ανταγωνισμό αυτό έχει να κάνει με την παραγωγή δεν μπορούμε να πετύχουμε μεγέθυνση της οικονομίας μας και δεν μπορούμε να έχουμε επομένω ε, τις οικονομίες κλίμακας όπως οι Αμερικανοί οπότε και μέσα από αυτές τις διαπιστώσεις ανεδίθη η Λευκή Βίβλος του Ζακ Ντελόρ ε, οι αναλύσεις της δεκαετίας του 80 και γι' αυτό και έγινε και η κατάργηση ένα σωρό φραγμών μη δασμολογικών. Είχαμε την ενιαία αγορά, είχαμε τις τέσσερις ε, βασικές ελευθερίες διακίνησης και έτσι απελευθερώσαμε, έτσι προχωρήσαμε στην νομισματική ολοκλήρωση και παρά ε, αυτές τις σημαντικές προόδους για την οικονομική ολοκλήρωση και παρά το γεγονός ότι αυτά έγιναν στη δεκαετία του 90 μέχρι αρχέ της δεκαετίας του 2000 και είχαμε τις πιο μεγάλες τότε συγχωνεύσει και εξαγορές ε, ρεκόρ στην οικονομική ιστορία και γι' αυτό τον λόγο α, ε, ανεδίθησαν και κάποιοι γίγαντες της εμπορίας και της βιομηχανίας χημεία, αυτοκινητοβιομηχανία ε, αυτές μπορούν να συγκριθούν με κάποιες αμερικανικές, αλλά συνολικά δεν μπορούν να συγκριθούν με την Αμερική. Επομένω, πρόκειται για μια ολοκλήρωση προχωρημένη και πλευρά τεχνολογική ε, συνέχισε να έχει η Αμερική καλύτερε επιδόσει. Παρά επομένω ε, το ενιαίο νόμισμα, την ενιαία αγορά, η Αμερική είχε μια ανάπτυξη η οποία βασίστηκε περισσότερο στην τεχνολογία, στην πληροφορία και ελάμβαναν υπόψη περισσότερο τις δυνατότητες της παγκοσμιοποίηση, της διεθνοποίηση της παραγωγής και χρησιμοποιούσαν τις αναδυομένες χώρες για να οργανώσουν την παραγωγή τους. Και επικεντρώθηκαν ε, περισσότερο οι Αμερικανοί στην έρευνα και ανάπτυξη. Και σε αυτό που λέμε branding. Στη δυνατότητα δηλαδή να φτιάξουν κάποιες, κάποιες επωνυμίες, κάποια σήματα παγκοσμίου κύρους. Οπότε εστράφησαν προς τις ε, ε, αναδειωμένες χώρες, χρησιμοποίησαν την Αλένα στην Νότια Αμερική, επίσης και την ε, Νότια Ασία, οργανώθηκαν στα δίκτυα παραγωγής και ε, αυτό αφορούσε κυρίως τον κλάδο της πληροφορικής. Apple, Microsoft και έκαναν, άρχισαν λοιπόν αυτή την υπεργολαβία που λέμε outsourcing προς ε, Ασία και τελικά και προς την Κίνα. Από το τέλος δεκαετίας του 1990 ε, διαπιστώσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σημειώθηκε πρώτο για τις νέες τεχνολογίες, τις νέες οικονομίες και στην πληροφορική με αυτές τις νέες εταιρείες τους νέους τομείς και κλάδους που αφορούν το διαδίκτυο, την ε, τεχνολογία της επικοινωνίας, αλλά επίσης και σε νέους κλάδους όπως η νανοτεχνολογία και βιοτεχνολογία. Και εκεί οι Αμερικανοί ε, είχαν το πάνω χέρι από ό,τι φαίνεται. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είχαμε την σταδίκη της Λισαβόνας η οποία συνελήφθη και χαράχθηκε ούτως ώστε να μπορούσαμε να καλύψουν το χαμένο έδαφος ως προς τους Αμερικανούς στην έρευνα και την τεχνολογία διότι διαπιστώθηκε ότι σε κάποιο σημείο είχαμε τους Αμερικανούς οι οποίοι επένδυαν πάνω από το 0,8, ενώ 0,1% του ΑΕΠ στην τεχνολογία και στην έρευνα, στην πληροφορική και σε νέες τεχνολογίες γενικότερα. Πάντως το δικό μας το πλεονίτημα ήταν κάποιες άλλες πιο προδοσιακές βιομηχανίες όπως ε, αυτοκινητοβιομηχανία, χημεία, αλλά αυτές δεν είναι νέες τεχνολογίες, έχουν ηλικία ενός αιώνα. Οι Αμερικανοί όμως τις πραγματικά νέες ε, τεχνολογίες προχωρούσαν, οπότε και εμείς θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε το χαμένο έδαφος σε αυτούς τους νέους τομείς. Οπότε είχαμε και αυτή την, ε, την πρώτη Αμερικανική, αλλά είχαμε και τις αναδυόμενες ε, οικονομίες, γιατί στο, δεκαετία του 90, στον τρίτο κόσμο, είχαμε σε πολλές χώρες εξελίξεις και όσον αφορά το χρέος τους, το παραδοσιακό, αλλά άνοιξαν οι οικονομίες τους όσον αφορά τις ε, επενδύσεις από το εξωτερικό και αυτές οι χώρες έγιναν αυτό που λέμε ασιατικός τίγρης. Αλλά έχουν βέβαια και την Ιρλανδία. Οπότε ανοίξανε προς τους επενδυτές, προς τις ε, πολυεθνικές και άρχισαν να γίνονται ζώνες ε, μονταρίσματος. Οπότε είχαμε και αυτές τις έμεσες συνέπειες, το spillover, ε, το, γιατί άρχισε να αγγίζει η τεχνολογία αυτή η Τουρκία, Ταϊλάνδη και Κίνα. Οπότε άρχισαν αυτές οι χώρες να συμμετέχουν σε αυτά τα δίκτυα των, της Ευρώπης, ε, της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και είχαμε όμως και τις τοπικές βιομηχανίες που μπορούσαν να, ε, να βγουν στην διεθνή εμπορική σκηνή και να ασκήσουν τον δεσμό. Samsung, Acer, Νότια Κορέα, Κίνα, Γιαγουάη και αυτές τελικά γίνανε ε, πολυεθνικές. Στη δεκαετία του 2000 αντιλαμβάνεται η Ευρώπη και βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις αναδυόμενες χώρες ικανές να εξάγουν ε, μεταποιημένα προϊόντα με τεχνολογικό περιεχόμενο ακόμα και αν εκείνε δεν ελέγχουν όλη τη διαδικασία παραγωγή στην τεχνολογία, αλλά εκείνε κάνουν τι εξαγωγέ τουλάχιστον. Και από την άλλη πλευρά, οι αμερικανικέ εταιρείε, οι οποίε είναι εντατικέ τεχνολογικά και είναι ικανέ να διαχειριστούν αυτά τα διεθνή δίκτυα παραγωγή, κυρίω του νέου τεχνολογικού κλάδου, με επιχειρήσει όπω την Microsoft ή την Apple. Συνεπώ, η στρατηγική τη Λισαβόνα έχει σαν αντικείμενο να κάνει την πιο ανταγωνιστική οικονομία, ανεβάζοντας το χρονολογικό επίπεδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προσπαθώντας να καλύψει αυτό το κενό ε, με τις ΗΠΑ και καθιστώντας πιο ευέλικτες αγορές εργασίας για να ευνοήσει ε, τις μεταφορές εργατικών, ε, εργατικού δυναμικού από τους φθήνοντες τομείς προς τους ακμάζοντες τομείς για να μην χάσουν τα ανταγωνιστικά τους πλέον εκτήματα οι Ευρωπαίοι με τις αναδυόμενες χώρες και να μπορέσουν να αγγίξουν αυτές τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης. Αυτές οι, αυτή ήταν η στρατηγική ε, της Δανίας, δηλαδή ε, το μοντέλο της Flexi Security, της ε, ασφάλειας και ελαστικότητας, με, που με τον Επίτροπο της εποχής προσπάθησε να δείξει ότι αυτή η στρατηγική επιτρέπει μεγάλη ευελιξία και ευνοεί το πέρασμα από ένα εργατικό δυναμικό το οποίο θα έχει μεγαλύτερα προσόντα ε, Περνώντα από του φθήνοντε τομεί προ του ακμάλλοντε τεχνολογικά τομείς, δηλαδή ε, τους τομείς τεχνολογίας πληροφόρησης. Επίσης, ε, να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τι ικανότητε τους για να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το κενό. Λοιπόν, η Στατική Λισαβόνα χρησιμοποίησε αυτό το αμερικανικό μοντέλο όπου οι εταιρείε εξειδικεύονται στου τομεί τη τεχνολογία, έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και φετέρου το branding, δηλαδή δηλαδή την ικανότητα δημιουργίας brands, δηλαδή εμπορικών ονομασιών όπως το Windows, το Apple, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά ε, αυτή η ικανότητα τεχνολογικής καινοτομίας ε, επιβάλλει νέες τεχνολογικές προδιαγραφές όπως κάνει η Microsoft με το Windows, όπως η Apple ή η Samsung και αυτή η ικανότητα καινοτομία δημιουργεί νέα τεχνολογικά πρότυπα ε, στη διεθνή αγορά αλλά και η ικανότητα να υπάρχει branding, δηλαδή ε, μια εμπορική ονομασία γνωστή διεθνώς ώστε οι πολυεθνικές να ελέγχουν τα διεθνή δίκτυα παραγωγής. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο. Η στατική της λοιπόν προβάλλεται σε αυτά τα πλαίσια με αυτό το στόχο, δηλαδή να υπάρχει η οικονομία της γνώσης και η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου. Φυσικά αυτός είναι ένας στόχος, ο οποίος ήταν υπερβολικά φιλόδοξος πιστεύω και κυρίως χωρίς να προβάλλει μία σαφή στρατηγική και τακτικές σαφείς για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων μέσα σε μια δεκαετία. Το πρώτο λοιπόν το οποίο μπορούμε να πούμε για τη στρατηγική Λισαβόνας και δεν θέλω τώρα να επισέλθω σε όλα, σε όλα τα έγγραφα που υπάρχουν, εκθέσεις του 2005, γνωρίζετε πολύ καλά ότι επικρίθηκε αυτή η ανοιχτή συντονιστική μέθοδος ως μία μέθοδος όχι πολύ δεσμευτική. Ε, λέχθη ότι υπάρχουν πολλοί στόχοι και ότι η Lisbon Strategy, η στρατηγική της Λισαβόνας αφορούσε τα πάντα και τίποτα αναφέρθηκε ότι τελικά δεν υπήρχαν ε, ποσοτικοποιημένοι στόχοι, όχι σαφείς και συνεπώς Εάν άλλοι δεν πραγματοποιούσαν αυτό το στόχο, τότε και εμείς δεν έπρεπε να το κάνουμε. Και συνεπώς είδαμε σε αυτές τις μεθόδους πολλές αδυναμίες στον τρόπο όπου δεν υπήρχαν δεσμευτικά κριτήρια, δεν υπήρχε υπερηθνικός έλεγχος, υπήρχε μόνο διακυβερνητική διάσταση και προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε μια στρατηγική που δεν ήταν διαφορετική, ενώ τα επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης των κρατών μελών διέφεραν πολύ. Αν δούμε εδώ την κατάσταση ε, βλέπετε ότι τη στιγμή που αρχίζει η στρατηγική της Λισαβόνας, ποια είναι η σύγκριση μεταξύ Ρουμανίας που ξοδεύει 0,4 του ΑΕΠ της και η Φιλανδία που ξεπερνάει το 3. Δηλαδή ένα επίπεδο που μπορεί να συγκριθεί με την Νότια Κορέα και τη Ιαπωνία το να πούμε ότι θα ακολουθούσαν την ίδια ταχύτητα ανάπτυξης ε, όσον αφορά τις γνώσεις αυτές οι δύο χώρες ε, δεν ήταν σωστό παρά το γεγονός ότι οι στόχοι ήταν εντελώς διαφορετικοί. Κάπου όμως υπάρχει μια έλλειψη ομοιογένειας, ετερογένεια πολύ μεγάλη. Από αυτή την άποψη πιστεύω λοιπόν ότι το βασικό σφάλμα είναι ότι δεν είδαμε ακριβώς τη μεγάλη τερογένεια που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών και αυτό το υπάρχει ε, τα business clusters, η, τα σύνολα, τα βιομηχανικά. Βλέπουμε τις νέες θεωρίες της διεθνούς οικονομικής γεωγραφίας, ότι δηλαδή τελικά υπάρχουν αυτά τα ε, clusters, τα βιομηχανικά clusters, έχουμε ε, ε, στην Μασαχουσέτη ή στην Καλιφόρνια τέτοια mm. παραδείγματα, δηλαδή μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση βιομηχανιών στον ίδιο τομέα. Και αυτή η στην καλιφορνια τετοια παραδειγματα δηλαδη μια πολυ μεγαλη συγκεντρωση βιομηχανιων στον ιδιο τομεα και αυτη η συγκεντρωση των βιομηχανιών δημιουργεί εξωτερικές οικονομίες κλίμακο που ωφελούν όλο αυτό το business cluster και του επιτρέπει να προσελκύσουν ε, το εργατικό δυναμικό με τα περισσότερα προσόντα και φθηνά. Τη στιγμή λοιπόν που έχετε αυτά τα αυτά τα φαινόμενα υπάρχει έλλειψη ομοιογένεια μεταξύ των χωρών που έχουν αυτά τα προσόντα και εκείνων που δεν έχουν. Διότι μπορούμε να πούμε ότι σε αυτού του τομεί διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οικονομίες κλίμακας στην έρευνα και την ανάπτυξη ακριβώς και η τεχνολογική πρόοδος των γεωγραφικών ζωνών που έχουν αυτά τα προσόντα ε, διαφέρει σε σχέση με εκείνες που δεν διαθέτουν αυτά τα προσόντα. Αυτό δεν είναι φαινόμενο που αφορά μόνο την Ευρώπη. Και στην Νότια Κορέα υπάρχουν τέτοιες ε, ανεπτυγμένες περιοχές, στην Σεούλ για παράδειγμα και άλλες περιοχές της Κορέας, της Νότιας Κορέας είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. Το ίδιο βλέπουμε ε, όπως στην Αμερική, η Λουιζιάννα, ή άλλες περιοχές Αμερικής. Καλιφόρνια, για παράδειγμα, έχουν πολύ αναπτυγμένη τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε μια ομοσπονδιακή χώρα, δεν είναι μια ενιαία χώρα και υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που είχαν πολλά προσόντα τεχνολογικά, όπως στην ορισμένε περιοχές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Σκανδιναβικών χωρών, της Γαλλίας και άλλες χώρες οι οποίες δεν είχαν αρκετά ανεπτυγμένη τεχνολογία η Roumanie. il y a des districts marsaliens, mais c'est dans l'industrie du textile et de certains assemblages. Vous avez des... Υπάρχουν euh, ε, μεγάλες ανεπτυγμένες περιοχές στη Σλοβακία όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Mm. Αλλά ήταν πολύ επικεντρωμένες αυτές τις τεχνολογίες στην βόρειο-δυτική Ευρώπη και ακόμα και μέσα στις χώρες δεν υπάρχει ομοιογένεια. Αν πάρετε για παράδειγμα την ε, περιοχή του Λονδίνου είναι πολύ πιο προηγμένη από ότι το ε, υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Και συνεπώς υπάρχουν ορισμένε περιοχές Marshall ε, που αφορούν αυτές τις χώρες. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που δεν έχουν καθόλου ανεπτυγμένες ζώνες στην τεχνολογία πληροφόρησης στις νέες τεχνολογίες, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία. Αυτό συμβαίνει και στην Νότια Κορέα και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Φυσικά, η ετερογένεια στι ΗΠΑ μπορεί να διορθωθεί με μεταφορές που γίνονται από τη μία πολιτεία στην άλλη, ε, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λόγω ε, της αδυναμίας των υπερεθνικών προπολογισμών και την έλλειψη των μηχανισμών. Συνεπώς, η στρατηγική της Λισαβόνα διαμορφώθηκε χωρίς να οργανωθούν μεταφορές και χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι εάν έχετε συγχρόνως μία βελτίωση της ευρωπαϊκής Ενσωμάτωση με ελευθερία κυκλοφορία του, του εργατικού δυναμικού και του κεφαλαίου, αλλά χωρίς στρατηγική για να δημιουργηθούν ε, πολύ ισχυροί πόλοι, ε, υπό τον Μπρίντον, υπό τον Μπάγκερμαν, ε, μπορούσαν τότε να, να προωθήσουν μια πολιτική ανταγωνισμού και να δημιουργήσουν μια κάθετη βιομηχανική πολιτική σε σχέση με τις οριζόντιες πολιτικές που δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτούς τους πόλους, τους ισχυρούς ε, ε τεχνολογικά πόλους, δημιουργήθηκε ένας χώρος πολύ ρευστός, οικονομικός χώρες ε, ρευστός και μπορούσαν οι χώρες να προβάλλουν την παραγωγή τους ανάμεσα με τα συγκριτικά πλεονέκτημα που είχαν, όπου όμως οι πολυεθνικές αποφάσισαν να επικεντρώσουν την έρευνα και την ανάπτυξη εκεί όπου υπήρχαν ήδη αυτοί οι ισχυροί πόλοι και να επικεντρώσουν τις δραστηριότητες του συναρμολόγησης που σε ορισμένε χώρε που, της τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και ήταν πιο ευέλικτο το εργατικό δυναμικό υπήρξαν χώρες μέσα σε αυτή την χαίρεση της εργασίας, την κατανομή της εργασίας, που γνώρισαν ειδικεύσει που δεν ήταν πολύ ευνοϊκές για τη χώρα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ 2000 και 2010 οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κατέδειξαν ότι τελικά η στατική της Λισαβόνας δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτές τις χώρες. Οι χώρες ε, του νότου της Ευρώπης, μπορούμε να ονομάσουμε την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία για παράδειγμα, και η Ιταλία όμως το ίδιο, ορισμένες λοιπόν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επίσης, και εδώ πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση, υπάρχει διαφορά μεταξύ των χωρών όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, που έχουν πολύ χαμηλή πρόοδο και άλλες χώρες όπως η Εσθονία και η Τσεχική Δημοκρατία που έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Βλέπουμε όμως ότι δημιουργείται μια μεγάλη, ένα μεγάλο τεχνολογικό χάσμα σε αυτή τη δεκαετία με φαινόμενα από βιομηχάνηση σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και αναδιοργάνωση αυτής της βιομηχανοποίηση προς ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που θα εξειδικευθούν στην συναρμολόγηση ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων. Αυτή η στρατηγική της Λισαβόνας λοιπόν δεν μπόρεσε να δει ε, πώς θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτές οι χώρες που εξειδικεύτηκαν και που δεν αναπτύχθηκαν αρκετά τεχνολογικά, εξειδικεύθηκαν στον τουρισμό για παράδειγμα, στις κατασκευές ή στη διεύρυνση του δημόσιου τομέα όπως είδαμε στην Ελλάδα. Και δεν επιμείναμε στο γεγονός ότι αυτές οι χώρες, καθώς προχωρούσαμε στο χρόνο, αυτές οι χώρες δεν είχαν καλές επιδόσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εδώ Βλέπετε στις διαφάνειες που σας έδωσα αυτό το τεχνολογικό χάσμα. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας και της ανάπτυξης της Eurostat που βλέπετε εδώ, αυτό το διάγραμμα το οποίο έφτιαξε η εταιρεία Πατέλ είναι ένα πολύ σαφέ διάγραμμα, το οποίο μας δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ετερογένεια ε, ανάμεσα στι χώρες, για παράδειγμα τη Φιλανδία φαινό και τη Ρουμανία φετέρου. η Φιλανδία και η Σουηδία συγκαταλέγονται μεταξύ των πολύ προηγουμένων χωρών, ενώ ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ είναι και η Ιταλία, όχι μόνο η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, αλλά και η Ιταλία είναι χώρε που δεν έχουν προχωρήσει αρκετά, όχι πιο πολύ από την Κίνα και λιγότερα προχωρημένε από ότι οι αναδυόμενε οικονομίε, όπως η Ταϊουάν ή η Νότια Κορέα. Συνεπώς, Υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες που δεν έχουν μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη νέα κατανομή της διεθνή κατανομή εργασίας και δεν μπορούν να ελέγχουν τα διεθνή δίκτυα παραγωγής όσο αποτελεσματικά το κάνουν οι αμερικανικές, οι ιαπωνέζικες βιομηχανίες και δεν είναι ανταγωνιστικές όσον αφορά την ευελιξία της εργασίας όπως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ή εκείνες που έχουν φθηνό εργατικό δυναμικό όπως η Τουρκία που μπορεί να συγκριθεί. Που, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα τη Ρουμανία και τη Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, η οποία σήμερα εξάγει ένα μεγάλο ποσοστό μεταποιημένων προϊόντων και σήμερα η Τουρκία είναι ικανή να, να δεχθεί κέντρα έρευνα και ανάπτυξη στην αυτοκινητοβιομηχανία με ευέλικτο εργατικό δυναμικό και χαμηλού μισθού. Το 55% του εργατικού δυναμικού στην Τουρκία. Ε, έχει, είναι χαμηλού κόστου, μεγάλη ευελιξία, πολύ μεγαλύτερη από την Ρουμανία και την Ελλάδα. Σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτέ οι χώρε θα μπορέσουν να βρουν τη θέση του στην παγκόσμια κατανομή εργασία σε μια οικονομία όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ αναδειωμένων χωρών που προσπαθούν να φτάσουν στι προηγουμένε χώρες και τις πολύ αναπτυγμένε χώρες όπως η Αμερική, οι σκανδινικές χώρες, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα που μπορούν να εξειδικευτούν στην οικονομία της γνώσης και την καινοτομία. Από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας στο να μειώσει το χάσμα. Εκείνο το οποίο είναι ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν φαίνεται να έχει λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2009 και τις επιπτώσεις που θα έχει όσον αφορά τη διεύρυνση του χάσματο μεταξύ των χωρών τη περιφέρειας που θίγονται περισσότερο από την κρίση και τι χώρε τη Βόρειας Ευρώπη που ανθίστανται καλύτερα στην κρίση λόγω τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση τη δομή των εξαγωγών του και τη τεχνολογική του δομή. Συνεπώ υπάρχει φόβο μέσα από τι πολιτικέ λιτότητε που υπάρχουν στι χώρε, όχι μόνο τη Ευρωζώνη, του νότου τη Ευρωζώνη, αλλά και στι χώρε τη περιφέρεια, όπω η Λετωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία. Υπάρχει φόβο λοιπόν να δούμε φαινόμενα brain drain, ε, αφέμαξης δηλαδή των εγκεφάλων, δηλαδή ε, να εξαγωγών των ικανών ε, από τη Ρουμανία και την Ελλάδα, οι οποίοι θα πάνε σε χώρες πιο ανεπτυγμένες, με μεγαλύτερους μισθούς, στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα όμως και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες οικονομίες, οι οποίες είναι πιο ισχυρές από τις δικές τους οικονομίες, τις προβληματικές. Λοιπόν, η στρατηγική 2020 όπως και η στρατηγική Λισαβόνας δεν ε, ε, δίνει μια λύση σε αυτό το τεχνολογικό χάσμα και δημιουργείται η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και να ρωτιόμαστε κατά πόσον η Νότια Ευρώπη θα γίνει το Μεξικό της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών όπως το Μεξικό είδαμε ε, ε, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το θέμα είναι αυτό μπορεί να συμβαδίζει με τις τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας, κυρίως την ελευθερία κυκλοφορίας του κρατικού δυναμικού. Βλέπουμε λοιπόν τις προστατευτικές λαϊκίστικες τάσεις ορισμένων οικονομικών ομάδων και πρωθυπουργών όπως ο Κάμερον που απροκάλυπτο αναφέρει στο Financial Times ότι η ελεύθερη διακίνηση στην Ευρώπη πρέπει να είναι λιγότερο ελεύθερη. Αυτό προέρχεται από αυτή την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και των χωρών της Περιφέρειας Ευρώπης. Αυτά ήθελα να σας πω. Είναι πολύ δύσκολο σε λίγα λεπτά να κάνει κανείς την, να την πλήρη εικόνα. Ευχαριστώ. merci beaucoup, monsieur Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεφρέν. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας ε, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κ. Λεβαντόφσκι. Σα ευχαριστώ. Εγώ ξέρετε ότι είμαι τακτικός επισκέπτης της Επιτροπής των Προπολογισμών. Λιγότερο στι δική σας, αλλά πάντως σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και πρόκειται για ιστορική συνάντηση. Η τελευταία συνεδρίαση αυτής της εντολής. Να σας πω ότι ο οργό προπολογισμό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σύμφωνα με τη στρατηγική τη Λισαβόνα και σύμφωνα με την ε, στρατηγική του 2020. Γιατί, σαν αφετηρία, είναι αυτό το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει. Γιατί πρόκειται για ένα από τα πολλά μα εργαλεία και ε, το οποίο βέβαια ε, είναι με τρίου βεληνικού, είναι 1% το ΕΠ και ίσω λιγότερο για την περίοδο 2010-2020. Και αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία των προπολογισμών έχουμε λιγότερα χρήματα από όλη την Ευρώπη για το μέλλον σε αυτή την περίοδο 2007 και 2013 μέχρι το 2013 και όπως είπαμε αυτό θα συζητήσουμε τώρα τι γίνεται με την στρατηγική της Λισαβόνας το στατική 2020 μετά να δούμε ποια είναι η συμβουλή του προπολισμού και να δούμε κάποιους σημαντικούς τομείς οι οποίοι ε, σαφώς συνάδουν προς αυτό το όραμα για την Ευρώπη του 2020. Ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη αξιολόγηση αυτής της στρατηγικής, κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2000 και ε, πηγή ήταν το ότι θα θέλαμε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ε, η Ευρώπη κάτω των προκλήσεων ε, του μοντέλου της Silicon Valley. Γιατί από εκεί κανείς μπορεί να καταλάβει Ποιο ήταν ο τρόπο ε, με τον οποίο οι Αμερικανοί μπόρεσαν να μετασχηματίσουν την οικονομία τους. Και έτσι μπορέσαμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες για την Ευρώπη και μιλούμε τώρα για τις προσπάθειες όλης της Ευρώπης, γιατί έχουμε και τις εθνικές προσπάθειες για να αποκτηθεί μια οικονομία βασισμένη στην ε, ε, γνώση. Καλά, να μην επαναλάβει ο καθηγητής Ντεφρέν για τις ε, αδυναμίες ε, και το δράμα που θα μπορούσε να ενεδρεύει το 2050. Κυρίως εμείς βλέπουμε τώρα το 2020 και θα πρέπει να δούμε το ότι σαν αδυναμία ότι δεν είχαμε θέσει κάποιες προτεραιότητες. Γιατί είναι πάρα πολλοί στόχοι και αυτό είναι κλασική περίπτωση ε, αδυναμίας. Δεν είναι επίσης σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ αρμοδιοτήτων εθνικών και ενωσιακών και θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο συντονισμός. Να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, εφαρμοστικός και εκτελεστικός. Να μην επαναλάβουμε σε αυτά που ελέγχθησαν, αλλά Θέλουμε μια στρατηγία το 2010 και θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι σε αυτή την περίοδο έχουμε 10 χώρες από τις 12 που μπήκαν, οι οποίες προέρχονται από την πρώην Σοβιτική Ένωση. Και αυτές οι χώρες δεν βρισκόντουσαν στο 60 του μέσου όρου του ενωσιακού, αλλά στο 30%. υπανάπτυκτες δηλαδή με αυτή την έννοια. Στρεβλής ανάπτυξης χώρες. γιατί όλες οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης αφορούσαν τον στρατιωτικό τομέα και όχι την οικονομία που έχει να κάνει με τον καταναλωτή. Οπότε και ήταν λάθος στρατηγική το να έχουμε μία στρατηγική για όλους. One size fits all αυτό το οποίο ίσχυσε την περίοδο 2000 έως 2004. Και όταν κάναμε την αναθεώρηση της Δίκης Λισαβόνας, συζητήσαμε τότε τη συμβολή του προϋπολογισμού και ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη την λισαβονοποίηση ούτως υπήν των διορθωτικών ταμείων που και αυτό είναι σημαντικό εργαλείο για να υποστηριχθεί αυτή η στρατηγική. Και αυτό έγινε με την δέσμευση κονδυλίων. Και το 60% των στόχων της ε, σύγκλησης θα πρέπει να καλύφθουν από την Λισαβόνα και 75% επίσης των στόχων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας. Οπότε έτσι να φροντίσουμε να γίνει η κατανομή των κονδυλίων. Οπότε και πετύχαμε κάποια πρόοδο. Ρίξω μια ματιά στο τι έγινε 2005-2007. Οπότε και είχαμε χιλιάδες με θέσεις αλλά κατόπιν ήρθε η χρηματοοικονομική κρίση σαν ράπισμα. τη στιγμή ακριβώ που είχαμε ευθυνη πολλά αποσχόμενη περίοδο 2005-2007 μετά την μεταρρύθμιση ΚΟΚ και την αναθεώρηση τη ε, στατική τη Λισαβόνα. Πάντω, πιο πολλά είναι τα δύνατα σημεία παρά τα πλέον εκτίματα σε αυτή την περίοδο. Πάμε τώρα στην φάση κατά την οποία θα πρέπει να δούμε κάποια συμπεράσματα. Μιλούμε για την περίοδο αυτή, του ενός του 2010 και μετά. Τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε αυτή τη νέα στρατηγική, αλλά όπως είπαμε η κρίση επισκέσει όλες αυτές τις προσπάθειες και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όταν κανείς έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση δεν μπορεί να έχει κατά το τι θα γίνει το 2020. Κανείς το 11 και το 12 δεν είχε κατά νου το τι θα γίνει το 2020. Όσοι λέγανε κάτι να γίνει, κάποια παρέμβαση για Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο κάτσαμε και σκεφτήκαμε πώς μπορούμε στο μέλλον να αντισταθούμε περισσότερο σε τέτοιες κρίσεις. Άρα αυτό, η αντιμετώπιση δηλαδή της κρίσης, ήταν το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση. Αυτό πρετάνευσε στην διαχείριση του προπολογισμού. Και ακριβώς αυτό που είχε ανάγκη η Ελλάδα το 2011 ήταν ο επαναπρογραμματισμός. Ήταν κάτι να γίνει με την, με την έλλειψη πιστώσεων, το credit crunch και όχι το τι θα γίνει το 2020. Οπότε και εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, αυτόν τον επαναπρογραμματισμό το front loading, την, την ενεργεία των νέων, αλλά όχι με ορίζοντα το 2020. Το πώς θα μπορούσαμε να χειριστούμε τα εργαλεία του προπολογισμού τότε, μέσα στην κρίση. Οπότε απαιτήθηκε διαχείριση και διακυβέρνηση στη στιβαρή από πλευράς του Συμβουλίου. Χρειάστηκε εντατική ε, προσπάθεια συντονισμού. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους μας. Και βέβαια να δούμε πώς θα αφιερωμίσουμε τον προϋπολογισμό με την στρατηγική του 2020. Πώς αυτός ο μικρός προϋπολογισμός θα γίνει καταλήτης πρόοδου. Να μην σταθούμε περισσότερο στα συμπεράσματα. Να δούμε κάποια γραφήματα, γραφικές παραστάσεις. Και πώς η αξιολόγηση θα βασίζεται στις επιτευχθεί επιδόσεις. Κάποια ξεκάθαρα κριτήρια τα οποία θα μας ε, βοηθήσουν να δούμε κατά πόσον στα πλαίσια της Αττικής 2020 σημειώνονται βήματα πρόοδου. Βέβαια πρόκειται εδώ για κάποιο είδους ε, ε, μακροοικονομικά κριτήρια τα οποία δεν είναι καθόλου δημοφιλή. Και αυτά τα βήματα γίνανε σε συνδυασμό με το Κοινοβούλιο και για τις νέες πρόπτικες και για τη στρατηγική 2020. Και είπαμε ότι ακριβώς με τέτοιους αξιολόγους θα πρέπει να ανοιχθεί η καλή απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινωνικών κονδυλίων. Βλέπετε τώρα σε αυτή την γραφική παράσταση ότι έχουμε έναν προπολογισμό που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας και μεταξύ του 2007-2020 έχουμε 32,3% ένα ποσοστό κονδυλίων το οποίο ακριβώς ανταποκρίνεται στους στόχους της στρατικής της Λισαβόνας. ανταγωνιστικό ε, κεφάλαιο 1α, 1β, συνοχή και στη συνέχεια για την γεωργία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοήσαμε τα άλλα κεφάλαια του προπολογισμού γιατί υπήρχε για Συρία και Ουκρανία πάρα πολύ μεγάλη πίεση να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια εσωτερικά δικαιοσύνη, πίεση και από το Κοινοβούλιο, το, τα οποία γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικά. Όμως, η συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τους στόχους της Λισαβόνας ήταν 30% μεταξύ 2007-2020 και έχουμε το 43,3% μεταξύ 2011 και 2013. Ανέβηκε δηλαδή. Και τώρα, από το 2014 και μετά έχουμε πάνω το 50%. για τους στόχους του 2020. Αλλά στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 πάμε στο 59% συμμόρφωση. Ξεκινούμε από έρευνα, πάμε σε ε, παιδεία, έρευνα, από τα κεφαλαία α α1β και για την γεωργία έχουμε όλο ένα και περισσότερη συμμόρφωση και υπαγωγή των προϋπολογισμών στην ε, συνθήκη και πολιτική της Λισαβόνης. Και τώρα, για να μπούμε στην τελική ευθεία αυτής της ε, ψυχικής μου. Βλέπετε εδώ ότι έρευνα και ανάπτυξη ε, χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία σαν τμήμα του προπολογισμού γιατί είναι τμήμα το οποίο αναπτύσσεται και είδαμε ότι έχουμε μετρέχουσες τιμές 80 δις όσον αφορά συγκρίσιμες τιμές 2007-2014 και βλέπετε ότι όλα αυτά τώρα ε, είναι ολοκληρωμένα στοιχεία και υπάρχει πρόοδος αλλά βλέπετε ότι εδώ πέρα οι δημόσιες δαπάνες φέρνουν καινοτομία αλλά έχουμε πάρα πολλέ διαστάσεις σε μια οικονομία της καινοτομίας, κάτι το οποίο ξεπερνά το τι κάνει δημοσίος τομέας, γιατί έχουμε και την επιχειρηματικότητα, έχουμε τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, έχουμε πάρα, πολλά, ε, πάρα πολλές επιμέρους υπόψεις ε, του θέματος που αφορούν αυτού τους τις δαπάνες. Αλλά όσον αφορά τον προπολογισμό, βλέπετε ότι σύμφωνα με τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου ανέβηκε η δαπάνη για ε, την έρευνα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον σφαιρικό ορίζοντα που καλύπτει μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από αποτελεσματική χρήση των πόρων όπως τα, την προσπάθεια προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση αλλά και την ε, προσαρμογή στον ψηφιακό κόσμο. Τώρα βλέπετε για τις υποδομές 2007-2013, ποιες είναι οι δαπάνες, εξυγχρονισμός των ε, υποδομών, είχαμε 8 δις, τώρα έχουμε 33,3, κυρίως για μεταφορές, μόχλευση του ιδιωτικού κεφαλαίου, τόσο ώστε να καλυφθούμε των κινδύνων για μακρόπνοα έργα και προγράμματα και για τα ενεργειακά 5,9, για τηλεπικοινωνίες και ψηφιακά επίσης. Παρ' αυτά, Πρέπει να σας τονίσω ότι τώρα είμαι θα υποπίεση λόγω των γεγονότων ε, ε, από πλευράς ανατολικών συνόρων να κάνουμε front loading όσον αφορά το κόσμο και την απασχόληση των νέων, κάτι το οποίο έγινε ε, εις βάρος του backloading των έργων υποδομής στην ενεργειακή πολιτική. Επομένως μετακινούμε κονδύλια από υποδομές ενέργειας προς τα έργα 2014 και μετά για το κόσμο και την απασχόληση των νέων. Αλλά πρέπει τη διασύνδεση των ε, ε, ενεργειακών θυλάκων να την φροντίσουμε οπότε είμαι στα υποπίεση για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις νέες ανάγκες που τόσο υπάρξει μια πολιτική μας χρειάζεται περισσότερο από το front loading. Μίλαμε για το 2014-2020. Αυτά όσον αφορά το τι έχει γίνει με αυτά τα ομόλογα έργων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό και χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον. Μετά έχουμε την επένδυση στην οικονομία της γνώσης. Το έρασμος εξελίσσεται, μεγαλώνει ισόβια κατάρτιση, ανταλλαγές, καλά για το μέλλον. Είτε αυτό γίνεται αυτοδικαίως και αυτομάτως, είτε τέλος πάντων έτσι είμαστε πιο κοντά στους στόχους του 2020 έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για να δομηθεί έτσι ο προϋπολογισμός για την, την έρευνα, την ισοβία κατάρτιση Οπότε μιλάμε για αύξηση του έργου κατά 40%. Τέλος έχουμε την πολιτική συνοχή. Οπότε και έχουμε εδώ πέρα πάρα πολύ σαφή ευθυγράμμιση με τις ε, συμφωνίες τερικής σχέσης, conditionality και τέτοιες συμφωνίες, τόσο ώστε έχουμε τώρα πάνω από το 90% της πολιτικής συνοχής το οποίο έχει ευθυγραμμιστεί με αυτό το οποίο ε, είναι η στόχη του 2020. Έχουμε μειώσει επίσης το περιθώριο λιγμών των κρατών μελών για τις ε, κρατικές δαπάνες περιφέρειες και για την Ανατολική Ευρώπη βέβαια ε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ε, λιγμών γιατί εκεί είναι περισσότεροι οι στόχοι. Αλλά θα πρέπει κανείς στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης να ε, αποδείξει την συμμόρφωσή του προς ε, τους στόχους του 2020 οπότε και οι καταβληθήσεις προσπάθειες ε, αμείβονται αναλόγως για στα πλαίσια των εργαλείων που έχουμε για την πολιτική συνοχή και εδώ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και βέβαια σαφώς ο προπολογισμό μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργαλείο επιτύχηση των στόχων του 2020 αλλά σαφώς όλα αυτά σκιάστηκαν, ευάρυναν από τα όσα ε, επιτάσσει ή από τα όσα απαιτούνται να κάνουμε λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης. Τώρα πάντως, θα πρέπει να στείλουμε προσπαθίες μα περισσότερο σε κάποιου δυναμικές ανάγκες της Ευρώπη και να έχουμε μια φιλοσοφία και, και, και φιλοσοφική προπολογισμού που θα αποκρίνεται στο μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα λοιπόν ε, ακούσαμε τις ε, δύο αυτές ε, ομιλίες και τώρα προβλέπεται το στάδιο των ερωταπαντήσεων και έχουμε κερδίσει και κάποιο χρόνο. Θέλω λοιπόν ότι τους αδέλφους, αν θέλουν να αποβάλουν μια ερώτηση. Κυρία Γκρέσλε, ε, πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες ε, και με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Έχω μια ερώτηση και προς τους δύο. Παρουσιάσατε και οι δύο με εντυπωσιακό τρόπο πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ερωτώ, χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Εστονία, η Γαλλία, τι θα συμβουλεύατε τις χώρες αυτές. Και νομίζω ότι δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα χρήματα. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις δυνατότητες που έχουν επιχειρήσεις. Είπατε και μόνοι σας πόσο μεγάλη είναι η σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών ε, και της επιχειρηματικής τους ε, πολιτικής. Πώς πρέπει λοιπόν να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επιχειρηματική πολιτική έτσι ώστε τα κονδύλια που διατίθενται να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Νομίζω ότι αυτή η ακρόαση είναι πολύ σημαντική για μας γιατί σε μια κρίσιμη περίοδο βλέπουμε ε, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα λοιπόν τίθεται το ερώτημα κατά πόσον στο μέλλον θα είναι δυνατόν με την αξιολόγηση επιπτώσεων και με το τεστ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες καλοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Και δεύτερον πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τις υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης. Και το τρίτο και σημαντικότερο ερώτημα είναι το εξής, ε, ότι έχουμε ε, τις ε, δέκα σημαντικότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες είναι εκείνες όμως που καταστρέφουν την απασχόληση στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν νομοθετικές πράξεις που όχι μόνο παρεμποδίζουν αλλά και καταστρέφουν τις απασχόλησης. Θεωρείτε ότι στο μέλλον με μία impact assessment, μία αξιολόγηση επιπτώσεων αυτό θα μπορεί να καθίσταται περισσότερο σαφές. Ο κύριος Γιάν Μούλντεν. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και οι ερωτήσεις που ετέθησαν πολύ σημαντικές. Ε, αυτό που δεν άκουσα στις ομιλίες ε, είναι ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Βλέπουμε ότι μιλάμε για το 1 του 100, ε, μάλλον ε, το ποσοστό για, για την έρευνα από το ΑΕΠ είναι 3%. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα που να μπορούμε να προβάλλουμε στην κοινή γνώμη και να πούμε ότι να, αυτό επιτεύχθηκε χάρη της Ευρώπης γιατί αλλιώς δεν θα σημειώνεται επιτυχία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και εγώ έχω να υποβάλω ένα ερώτημα προς τον κύριο Ντεφέγκ. Συγκεκριμένα το εξής. <clears throat> Αναφερθήκατε στην ε, διαρροή εγκεφάλων και κατ' ουσίαν εδώ πρόκειται για ένα φαινόμενο που υπάρχει. Οι συνάδελφοι από τη Βουλγαρία αλλά και από άλλες χώρες επισημαίνουν ότι στη Βουλγαρία εκπαιδεύονται γιατροί, πληρώνονται από το βούλγαρο φορολογούμενο και τελικά πολλοί από αυτούς φεύγουν σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, την Ελβετία αλλά και στο Βέλγιο. Και αντίθετα πολλοί Γερμανοί πτυχιούχοι και αυτοί φεύγουν από τη Γερμανία, πάνε στην Νορβηγία, πάνε στην Ελβετία και κάτι άλλο. Ε, αν επισκεφτεί κανείς χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Ρουμανία, εγώ τις επισκέφτηκα πριν από 1,5 χρόνο με το ποδήλατο, κάναμε ένα τουρ στο Δούναβι ε, και αν ρωτήσει κανείς ε, νέους ανθρώπους εκεί σε αυτές τις χώρες το τι θα κάνουν λένε θα φύγω, θα πάω στο Λονδίνο, θα σπουδάσω πληροφορική θα πάω στο Μόναχο ή στην Καλστρούη και θα σπουδάσω μηχανολόγος και όταν τους πει κανείς μα μην εδώ γιατί δεν μένεις εδώ και λένε μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα εδώ γι' αυτό λοιπόν πείτε το ερώτημα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε αυτές τις χώρες και μπορούμε να τους πούμε να μην σπουδάσουν, να μην ενταχθούν και αυτοί στους, σε αυτή την πολιτική των ε, παγκόσμιων παικτών ή μήπως ε, θα πρέπει τέλος πάντων και αυτοί οι νέοι να έχουν μια διεθνή εκπαίδευση. Όμως το ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους κίνητρα θα υπάρχουν για αυτούς τους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν και επίσης ε, κατά πόσο ενδεχομένως θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο ορισμένα ερευνητικά ιδρύματα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα είδος πυρήνα ε, ο οποίος ε, πυρήνας θα μπορεί να επιτρέπει και τη μεταφορά τεχνολογίας. Σε σχέση λοιπόν αυτό το ερώτημα με το άλλο για την αφέμαξη των εγκεφάλων μπορούμε ίσως να πούμε ότι ίσως μετά από κάποια χρόνια να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη αυτής της μορφής γιατί και το Silicon Valley ε, με αυτόν τον τρόπο προέκυψε η Καλιφόρνια πριν από 100 χρόνια δεν ήταν αναπτυσσόμενη περιοχή τότε ήταν το Χάιο άλλες ε, χώρες, το Illinois Τώρα όμως φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτές και πάνε στην νέα βιομηχανία. Ε, δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει ο Επίτροπος ή ποιος θέλει να, να αρχίσει. Παρακαλώ. Thank you. I was expecting advice, not necessarily questions. <laughs> Κοιτάξτε, εγώ περίμενα να μου δώσετε συμβουλές, όχι να μου υποβάλλετε απαραίτητα ερωτήσεις και θέλω να πω το εξής. Το τελευταίο σας σχόλιο κατά κάποιον τρόπο σχετίζεται με τα σχόλια της κυρίας Κρέσλε. Δηλαδή, ε, στο κατά πόσο μπορεί να υπάρχει μία συνταγή για όλες τις χώρες. Εγώ δεν έχω, ίσως έχει ο συνάλφος ο κύριος Ντεφρά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί έχουμε κάποια εργαλεία ανάπτυξης στους ευρωπαϊκούς προπολογισμούς. Υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους, ας πούμε, από την Ανατολική Ευρώπη να αποκτήσουν καλύτερη εκπαίδευση, παραδείγματο χάρη στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Όμως ε, πρόκειται για ε, ένα δίκοπο μαχαίρι, μπορεί και να μην επιστρέψουν ποτέ. Το πρόγραμμα Έρασμος βοηθάει στο να κάνει κανείς ε, σταδιοδρομία σε μια άλλη περιοχή της Ευρώπης ε, με καλύτερες αμοιβέ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά τα προγράμματα. Νομίζω ότι μπορεί να προκύψει καθαρό όφελος ας πούμε για την Πολωνία αλλά δυστυχώς τέτοιου προγράμματα μπορούν να επιτείνουν και την ε, μετανάστευση. Στη Ρήγα, στη Λετωνία μου είπαν ότι να μην προωθήσουν τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα για τους νέους γιατί οι νέοι έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε μετακίνηση και ίσως ε, τελικά αυτοί ε, μετακινηθούν προς μία κατεύθυνση που δεν είναι εφικτή. Πρόκειται λοιπόν για ένα δίκοπο μαχαίρι όπως σας είπα και η απάντηση για τη σημερινή Ευρώπη δεν είναι ένα μέτρο που να ταιριάζει για όλους γιατί υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές νοοτροπίες και στους δημόσιους υπαλλήλου και στους βιομηχανικούς κύκλους. Ο κύριος Ρούμπιχ μετατόπισε λιγάκι το όλο θέμα από την καινοτομία στην απασχόληση και πολύ σωστά με τον τρόπο αυτό αναφέρθηκε και στις πολιτικές επιπτώσεις ε, της ανεργίας των νέων. Και πάλι λοιπόν εδώ υπάρχει ένα παράδοξο και θα μου επιτρέπετε να προκαλέσω λιγάκι. Όταν ε, έγινε μία μελέτη για τις επιπτώσεις των διαφόρων προγραμμάτων στην απασχόληση διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλύτεροι πολλαπλασιαστές είναι στην, στις υποδομές, όχι στην έρευνα και την ανάπτυξη. Και αυτό ε, φάνηκε σε αρκετές χώρες να σας πω παραδείγματο χάρη ε, πώ οι επενδύσει βοήθησαν τη δική μου τη χώρα, την Πολωνία, να αναπτυχθεί. Αλλά οι πολλαπλασιαστέ μερικέ φορέ βρίσκονται στι υποδομέ. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε ε, τέτοιου είδου προγράμματα. Η απασχόληση είναι εξίσου σημαντική σήμερα όπως και η οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Και τα δύο είναι απαραίτητα. Και όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, αυτή είναι μια κλασική ερώτηση που έχει σχέση με το σε ποιο βαθμό οι υπερβολικές αυτές διατάξεις παρεμποδίζουν κατά κάποιον τρόπο την ανάπτυξη της Ευρώπης. Για πρώτη φορά είμαι στην ευτυχή θέση να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακύρωσε μάλιστα κάποιους κανονισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την αρχή της επικουρικότητας και νομίζω ότι ε, μια πολύ σημαντική θέση στους επόμενους επιτρόπους, στην επόμενη επιτροπή θα είναι ο Επίτροπος για τις ε, νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ο κ. Μούλντερ ρώτησε σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε με τους ε, πόρους που διαθέτουμε. Και εδώ θέλω να σας πω ότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, τα 80 δις, αυτά θα πρέπει να υπολογίζεται και με βάση τη συγχρηματοδότηση. Στα ερευνητικά προγράμματα η δική μας συνεισφορά είναι το ίμιση. Το υπόλοιπο μισό προέρχεται από κίνητρα που ε, προσφέρονται από τη Μεγάλη Βρετανία ή από ερευνητικά κέντρα στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει η συγχρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στην έρευνα και την ανάπτυξη μπορούμε να ε, έχουμε δυνατότητα να προκαλέσουμε τις επενδύσεις και όσον αφορά τη συνοχή πράγματι εκεί η συγχρηματοδότηση είναι πολύ πιο περιορισμένη και ε, τα κίνητρα προσφοράς είναι πολύ πιο περιορισμένα. Αυτά είναι τα δικά μου τα σύντομα σχόλια. Ε, alors, je Λοιπόν, θα ήθελα να απαντήσω πρώτα σε εσά. Νομίζω ότι υπάρχει πράγματι μια διαφορά ε, στον τρόπο που στι ΗΠΑ ο ιδιωτικό τομέα ασχολούνται περισσότερο με την έρευνα και την ανάπτυξη και ιδιωτικέ ιδιωτικές επιχειρήσεις, αν θέλετε, έχουν σημαντικότερο ρόλο στην Αμερική από ό,τι στην Ευρώπη, το οποίο όμως συνδέεται και με την ανάπτυξη του venture capitalism, του καπιταλισμού κεφαλαίων κινδύνου. Όλες οι αναδυόμενες επιχειρήσεις, τι startups, δεν περνάνε από τους χρηματοοικονομικούς κύκλους από ό,τι στην Ευρώπη. Το venture capitalism στις startups στην Αμερική αφορά της ε, Silicon Valley ή το Want to Wait ε, στη Μασακουσέτη. Συνεπώς, σε αυτά τα πλαίσια έχουμε λιγότερο venture capitalism στις λιγότερο προηγμένες περιοχές στην Αμερική. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του venture capitalism που θα μειώσει αυτό το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών. Από αυτή την άποψη λοιπόν πιστεύω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το γεγονός ότι κρατημέλη έχουν μια περιφερειακή θέση όπου δεν υπάρχουν district μαρσαλιά, όπου δεν υπάρχει ευκολία στην πρόσβαση. Δηλαδή όσον αφορά τις υποδομές υπάρχουν χώρες περιφέρειας που, όπου πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση και δύσκολα μπορούν να ενταχθούν στα διεθνή δίκτυα παραγωγής και συνεπώς να δημιουργήσουν αυτές τις περιοχές δεν θα δημιουργήσετε district μαρσαλιά από το μηδέν. Η κινέζικη κυβέρνηση δημιουργεί τέτοιες περιοχές στην περιοχή του Σινγκ Στι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή πρόκειται για μια πολύ δραστήρια βιομηχανική πολιτική που ε, με ανακατανομή από τις πλούσιες περιοχές, τις πιο φτωχές περιοχές της Κίνας και εκεί υπάρχουν κρατικές επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχει το κράτος και συνεπώς διαθέτει τα μέσα για να δημιουργήσει εκ του μηδέν αυτά, αυτές τις ζώνες. Δεν νομίζω όμως ότι το venture capitalism θα προχωρήσει προς την Ελλάδα, Πορτογαλία, τη Ρουμανία ε, ε, και, ότι η ιδιωτικό τομέα θα αναπτυχθεί πολύ εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές. Το δεύτερο, Πιστεύω ότι πράγματι το θέμα τη της των εγκεφάλων του brain drain είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ακόμη και η κινέζικη κυβέρνηση που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή οι περισσότεροι Κινέζοι φοιτητέ ε, στο εξωτερικό δεν επανέρχονται στην Κίνα. Διότι θεωρούμε ότι τα δύο τρίτα εξ αυτών δεν επανέρχονται στην Κίνα και προσπαθούν να δικτυωθούν στις πιο προηγμένες χώρες, κυρίως στις ΗΠΑ. Συνεπώς το θέμα των retenees, πώς να κρατήσει κανείς αυτούς τους εγκεφάλους, αυτά τα μυαλά στη χώρα πίσω είναι περίπλοκο ακόμα και για την Κίνα που έχει district Μάρσαλιά, βιομηχανική πολιτική πολύ πιο αναπτυγμένη, ε, κέντρα αριστείας. Υπάρχουν λόγοι ε, που οφείλονται στο πολιτικό σύστημα και στο επίπεδο ζωή στην Κίνα και εξηγούν γιατί δεν επανέρχονται οι Κινέζοι που έκαναν σπουδέ στο εξωτερικό. Ε, πρέπει όμω να είμαστε ρεαλιστέ. Θα επανέλθετε σε μια Βουλγαρία ή μια Ρουμανία όπου υπάρχουν λιγότερα νοσοκομεία, λιγότεροι δρόμοι, λιγότερε δημόσιε υπηρεσίε, λιγότερε υπηρεσίε κοινή ωφελία ε, μετά από την ε, πολιτική λιτότητα και μεγαλύτερη αστάθεια αν έχετε πολλά προσόντα, δεν ξέρω αν θέλετε να επανέλθετε σε ένα κλίμα κοινωνικοπολιτικό τη περιφέρειας. Σήμερα δυστυχώ στην Ελλάδα ή τη Ρουμανία. Το θέμα είναι πώς μπορεί να προσελκύσει κανεί αυτά τα κεφα... αυτά... αυτούς τους αυτά τα μυαλά και θα πρέπει λοιπόν να συνδεθούν ε, στα δίκτυα τα ευρωπαϊκά μέσω υποδομών και αυτό είναι το θέμα της απασχόλησης βεβαίως του εργατικού δυναμικού. Φοβούμε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα με, τα περιορισμένα κεφάλαιά τους δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα προς το παρόν. Είμαι αρκετά απεσιόδοξη σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να προσελκύσει πάλι αυτά τα μυαλά. Αν πάρουμε το παράδειγμα της Καλιφόρνιας, είναι πολύ ενδιαφέρον, ιστορικά αν θέλετε το θίξατε κι εσείς. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιοχές όπως η Καλιφόρνια που ήταν λιγότερα ανεπτυγμένες ε, σε σχέση με το Σικάγο ή άλλες βιομηχανικές περιοχές. Αν δούμε όμως πώς θα αναπτύχθη η Καλιφόρνια, δεν είναι μόνο τα πορτοκάλια, αλλά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είδαμε σιγά αναπτυχθηκε η Καλιφόρνια είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ε, της ε, βιομηχανίας εξοπλισμών και το Silicon Valley αναπτύχθηκε με βοήθεια αυτά τα στρατηγικά προγράμματα στην Αμερική. Το διαδίκτυο είναι τη Αμερική που δημιουργήθηκε με χρήματα του Μοσπονδιακού κράτου για να δημιουργηθεί ένα σύστημα επικοινωνία για το ναυτικό τη Αμερική. Πολλέ καινοτομίε τη IBM και της Microsoft έγιναν στα στρατιωτικά πλαίσια, στα πλαίσια του Star Wars ή πρωτοβουλειών της ε, κυβέρνησης Ρίγκαν που ήταν μια βιομηχανική πολιτική όπου η πρωτοβουλειων της κυβερνηση ριγαν που ηταν μια οικονομία ξόδεψε πολλά χρήματα για στρατιωτικές δαπάνες, 4% του ΑΕΠ, σε μια οικονομία στρατιωτική high-tech, υψηλή τεχνολογία. Και αυτές οι εφαρμογές έγιναν και στον πολιτικό χώρο, όχι μόνο στον εξωστρατιωτικό. Συνεπώς αυτά έγιναν με βοήθεια υποστήριξη του κράτους και με βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε ότι η Ρουμανία έφνης θα γίνει σαν την Καλιφόρνια, εάν δεν έχει τη βοήθεια που είχε η Καλιφόρνια από το Αμερικανικό κράτο. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι το Αμερικανικό κράτο δεν παρεμβαίνει. Εδώ στην Ευρώπη δεν πιστεύω ότι οι προπολογισμοί τη στρατηγική τη Λισαβόνα είναι ανύπαρκτοι, αλλά είναι πολύ περιορισμένοι πιστεύω και ανεπαρκείς ώστε να δημιουργηθούν υποδομές που θα επιτρέψουν στις, στις χώρες περιφέρειας της Ευρώπης να επανενταχθούν περισσότερο στην ευρωπαϊκή οικονομία για να δημιουργηθεί κάπου να υπάρχουν κίνητρα ώστε να μην υπάρχει διαρροή των μυαλών. Ως οικονομολόγος δεν μπορώ να πιστεύω ότι χωρίς μεγαλύτερη μεταφορά υπερεθνική όλα αυτά θα επιτευχθούν. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, δεν θα μπορέσουμε σήμερα να βρούμε τη μία και μόνη αλήθεια, αλλά με πάση περιπτώσει πιστεύω ότι μπορούμε να ορίσουμε περαιτέρω πολιτικές και στόχους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Λεβαντόφσκι και τον κύριο Ντεφρέν για αυτές τις ε, ομιλίες τους και προτείνω να προχωρήσουμε ε, αμέσως. Ε, ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο προλαλήσαντες που ήρθαν στη συνάντησή μας. liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, επόμενο μιλητή σχετικά με την στρατηγική της Λισαβόνας. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και τον κύριο Παουλ Κόπλαντ από το Queen Mary του Λονδίνου. Κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Κόπλαντ, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας ε, και όταν ε, τακτοποιηθούν τα τεχνικά ε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε που μας δίνετε ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο για την στρατηγική της αγοράς. Ονομάζεται ε, αξιολογώντας τις επιτυχίες και κατανοώντας τις αποτυχίες της στρατηγικής αγοράς. Πρόκειται για ένα βιβλίο εκεί όπου έχουμε συλλέξει τις γνώμες από τους καλύτερους εμπειρογνώμενους για όλα αυτά και πρόκειται για την πρώτη τέτοια πανεπιστημιακή μελέτη που κάνει γνώμη μου που έχουμε καλύψει όλες τις στρατηγικές, τις πολιτικές που καλύπτει η συνθήκη της Λισαβόνας ε, απασχόληση, ε, περιθωρισμός κοινωνικός, ε, υγεία, έρευνα, ανάπτυξη, παιδεία, οικονομική διακυβέρνηση σε σχέση με την ΩΝΕ. Εμείς οι οποίοι είχαμε την εμπειρία του βιβλίου, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια περίληψη και θα πρέπει να δούμε μέχρι πού θα φτάσουν αυτά, αυτά τα συμπεράσματα και να δούμε όλες αυτές οι πληροφορίες, πώς έχουν εξελιχθεί από τότε που το βιβλίο εκδόθηκε. Για να μπορέσουμε να σας τα εξηγήσουμε, πρόκειται να χωρίσουμε στα δύο αυτή την παρουσίαση. Θα ξεκινήσω εγώ με μια αξιολόγηση του ευρύτερου τοπίου σε σχέση με τα πλέον εκτήματα, τα όρια της Αττικής της Λισαβόνας, να μπορούμε να τα καταλάβουμε και στη συνέχεια ο συνάδελφος, ο καθηγητής Κόπλαν, πρόκειται να σας εξηγήσει τις πολιτικές ε, καθέκαστον όσα καλύπτει αυτό το βιβλίο. Οπότε προσωπικά ξεκινώ εστάζοντας την προσοχή σε τρεις άξονες που θεωρώ ότι μπορεί να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια αξιολόγηση της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας. Πρώτα πρώτα, να καταλάβουμε και να αξιολογήσουμε της στρατηγική Λισαβόνα σαν ε, ένα διάλογο, μια διαλεκτική μάλλον. Γιατί εδώ έχουμε δύο βασικότερα ζητήματα. Το πρώτο είναι το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δίκιο να θεωρήσει ως υψίστη προτεραιότητα του 2000 την ανταγωνιστικότητα. Και το ίδιο να επαναλάβει το 2010. Βεβαίω, αυτή η μέρημνα για ανταγωνιστικότητα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον ενιαίο μηχανισμό ε, ισοτιμιών και με το ευρώ. Και επίσης ο εντοπισμός συγκεκριμένου θέματος, ούτως ώστε κανείς να ξεκινήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, είναι μια αξιόλογη ιδέα. Παρ' όλα αυτά, η απόλυτη αγωνιστικότητα συνολικά που αποτελεί το βασικό σημείο αφετηρίας. Είναι κάτι το οποίο δεν ποτέ ήταν και κατά μου ούτε τώρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως μερικοί νομίζουν. Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη σε κάποιες ανθρώπινες χώρες πολλές φορές θεωρείται ε, στοιχείο και απόδειξη για τέτοιες ε, σκέψεις. Αλλά από την άλλη μεριά τι έγινε, πώς κλείθηκε το ΑΕΠ τους σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ και την άλλη μεριά το ότι είχαμε απώλεια ε, ανταγωνιστικότητας δεν είναι ένα φαινόμενο ευθύγραμμα όπως πολλοί θεωρούν. Ας πούμε, έχουμε για τον... Ε, ε για τον μηχανισμό ε, τρεχουσών συναλλαγών κάτι το οποίο δεν συνάδει προς την κρίση. Αυτό το οποίο έγινε όμως τα τελευταία χρόνια είναι το εξή ότι διαπιστώθηκε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει μία απόκληση της πορείας της ανταγωνιστικότητας με τους στόχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι μέχρι ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη αγγίλες αγώνας αμέλησε την ιστορική διάσταση της ανταγωνιστικότητας. Εδώ η απάντηση είναι ναι, καταφατική. Οι αρχικές ε, αναφορές στην ανταγωνιστικότητα και στην συνοχή αντικαταστάθηκαν από μια σύλληψη της ανταγωνιστικότητας που βασίζεται σε μια αιώνια διαμάχη, ανταγωνισμό μεταξύ των μελών. Η λογική πάντως Μα οδηγεί στο ότι αυτό το οποίο κερδίσαμε στην τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι ενό μεγάλου βαθμού είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί αιωνίω να μα οδηγεί στο να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Και αυτή η διαλεκτική για να μπορέσει να έχει κάποια βάση σε επίπεδο άσκηση πολιτική και σε εθνικό και συνολικό επίπεδο θα πρέπει τα πράγματα να είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Θα πρέπει να έχουμε πιο δαπανηρέ πολιτικέ αντιστάθμισης σε εθνικό, σε τομεακό ή σε άλλο επίπεδο, ή περιφερειακό επίπεδο, όπου κάποιοι να είναι μοιραίοι χαμένοι. Επίσης, αυτή η ανταγωνιστικότητα, η πολιτική μόνο για περισσότερη ανταγωνιστικότητα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθείται και αποτελεί μια φαινάκι το ότι αυτό μπορεί να γίνει με αυτόματο πιλότο από μόνο του. Βεβαίω υπάρχει ένα υπαρκτό κίνδυνο, δηλαδή ότι πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια τη Ευρωπαϊκή Κοινωνία πρόκειται να αποξενωθούν να βρεθούν στο περιθώριο αυτή τη διαδικασία και πορεία ολοκλήρωση. Ένα δεύτερο άξονα τώρα που να χρησιμοποιήσουμε, τόσο ώστε να αξιολογήσουμε την ε, ε συνήθεια τη αγώνα, είναι να δούμε ποια είναι η αρχιτεκτονική τη διακυβέρνηση. Ένα από του πιο δύσκολου τομεί για να ζυγίσουμε την επιτυχία και την αποτυχία. Σίγουρα. Οι απαντήσεις πάντοτε δεν μπορούν να είναι αμερόληπτες. Εξαρτάται ο καθένας πώς βλέπει τις ε, ολοκληρωμένες πολιτικές. Ίσως εδώ θα βοηθήσει να σκεφτούμε τα εξής δύο. Πρώτον, η ανοιχτή εδώ συντονισμού που ήταν το, το βασικό όχημα επίτευξης σκοπών η Λισαβόνα και η Ευρώπη 2020 μα οδήγησε σε μια διαδικασία λήψη αποφάσεων ξεκάθαρη που να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά παράλληλα με την παραδοσιακή κοινωτική μέθοδο. Κάτι γνώμη μου. Το ερώτημα σίγουρα είναι, το, η απάντηση συγγνώμη, είναι σίγουρα αρνητική. Δεν έχουμε καταρχήν μια ενιαία μέθοδο ανοιχτού συντονισμού. Έχουμε απλώς ένα σύνολο διαφορετικού βαθμού ανάληψη δραστηριοτήτων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, σύνολο δεσμεύσεων των μελών διαφορετικών. Και κάποιοι στόχοι ε, αποτιμώνται ποσοτικά, άλλοι όχι. Οπότε, η συγκρισιμότητα της προόδου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι είναι δύσκολο ακριβώς να μετρήσει και να συγκρίνει τα διαφορετικά κριτήρια και στόχους. Ακριβώς λόγω της μεθόδου που θέλει, της μεθόδου των, των διαρκτικών αλλαγών που θέλει να επιφέρει στα κράτη-μέλη η Ευρώπη. Κάτι άλλο θα πρέπει τώρα επίσης να λάβουμε υπόψη όταν μετράμε την επιτυχία της Λισαβόνας είναι το να δούμε κατά πόσον η ίδια αυτή η στρατηγική επέδρασε σε άλλες αυτό ήδη συζητήθηκε από τους προλαλήσαντες. Και έχουμε στοιχεία σαφή ότι ολένα και περισσότερο είχαμε λισαβονοποίηση μια σειράς πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως των διορθωτικών ταμείων. Αυτό καταρχήν είναι καλό, αλλά η συνέργεια μεταξύ στόχων της Λισαβόνας και υπαρχουσών πολιτικών δεν είναι πάντοτε σαφής. Και γι' αυτό οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να συνδέσει δύο πολιτικές, κάποιες πολιτικές με τους στόχους της Λισαβόνας δεν οδηγείται πάντοτε σε επιτυχία. Ένας τρίτος και τελικός στόχος που θα πρέπει να υπόψη είναι να δούμε την Λισαβόνα, την ε, η στρατηγική 2020 σαν ένα σύνολο μετρήσιμων στόχων. Σε επίπεδο μακροοικονομικό μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα κριτήρια σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας ή την στρατηγική του 2020. Κάτι το οποίο να το έχουν όλα τα κρατημέλη πετύχει. Σε ένα άλλο επίπεδο πάντως, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ευρωζώνη, τότε είχαμε ίσω τις πιο σαφείς ενδείξεις των, αποτυχία και τη Αττική Λισαβόνα και του Ευρώπη 2020. Κυρίως όσον αφορά τους βασικούς μηχανισμούς. Όπως τον εκτό συντονισμό. Ε, να προσέξουμε τα εξή τρία. Πρώτον, η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την κρίση στην Ευρωζώνη σε κάποιο πρώιμο στάδιο. Ας πούμε την εκτροπή της ε, ελληνικής οικονομίας ή τη ε, ανισορροπή τη αυξανόμενη Ιρλανδία και Πορτογαλίας Αυτά δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά το 2010. Αυτά όλα βαθμία σορευόντουσαν επί πολλά έτη. Όμω, αν διαβάσετε τι κατευθυντήριε, που είναι η πρώτη προσπάθεια ε, και κατευθυνόμενης στρατηγικής, θα καταλάβετε ότι δεν υπήρχε δυναμική προσπάθεια ούτε από ε, πλευράς κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο μακρονομικός συντονισμός. Οπότε, πώς να διαπιστωθεί ότι μια τέτοια διαδικασία μεταρρύθμισης είχε συνέπειες στα κρατη για την παιδεία ή για την ε, καινοτομία ή για την έρευνα. Ένα δεύτερο, το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε και εδώ διαφωνώ με τους είναι ότι θα πρέπει να σκεφτείτε την ε, αιτιώδη σχέση. Από τη μια μεριά έχουμε την ε, αποτυχία Λισαβόνας και του Πρωτοβουλίου 2020 να και του σκοπούς και από την άλλη μεριά το εξάσωμα τη κρίση κάθε αυτό. Θεωρούμε ότι η ρίζα της κρίσης ήταν το ότι είχαμε απόκληση στην ε, ανταγωνιστικότητα μας των μελών. Σχεδόν πριν από 15 χρόνια η στατική Λισαβόνας έδωσε την υπόσχεση ότι θα κάνει την Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική οικονομία. Ξέρουμε όμως τώρα ότι με την Ευρωζώνη όλο ένα και περισσότερο χάνουμε στην ανταγωνιστικότητα. Η έκθεση ΚΟΚ υποσχέθηκε από 10 χρόνια απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι μεταξύ 2004 και 2012 η απασχόληση στην Ένωση συνολικά αυξήθηκε μόλις 1%. Την ίδια περίοδο η απασχόληση στην Ελλάδα έπεσε 10%. Στην Ιρλανδία 8% και η Ισπανία και η Πορτογαλία κατά 6%. Πριν από τρία χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Ευρώπη 2020, είχαμε υποσχέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και συρρήγνωση της στόχης, αλλά από το 2010 το ΑΕΠ της Ένωσης σωρευτικά αυξήθηκε το ΑΕΠ κατά 3,4% για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα το ελληνικό ΑΕΠ συρρυκνώθηκε κατά 23%. Το πορτογαλικό κατά 19,6%. Το ισπανικό 9,5% και το ελληνικό κατά 7%. Ίσως κάποιοι να ισχυριστούν ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι αντικειμενικά και μερόληπτα γιατί ε, έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση. Όμως αυτό που θέλουμε να πούμε ότι ακριβώς επειδή η στατική Λισαβόνα και 2020 απέτυχαν στους στόχους τους, γι' αυτό ξεκίνησε η κρίση. Άρα θα ήταν σωστό να πει κανεί ότι με κάποιο τρόπο η κρίση της Ευρωζώνης ε, θολώνει την εικόνα και το ότι η αντικειμενική πραγματικότητα έχει άλλος. Τέλος. να δούμε πώς χαράσεται η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Η ανοιχτή του συντονισμού ότι είναι η μόνη ρεαλιστική μέθοδος όσον αφορά τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οπότε είχαμε κάποιο συντονισμό ε, ε, εκουσίου χαρακτήρα διακυβερνητικού χαρακτήρα που θεωρήθηκε ότι αυτό είναι το τίμημα για να πετύχουμε αυτόν τον συντονισμό. Αυτό το 2000 ήταν σωστό, αλλά όχι σήμερα και σίγουρα δεν θα είναι σωστό το 2020, για το 2020 ή τέλο πάντων όταν ε, αποφασίστηκε η τελο παντων οταν ε αποφασιστηκε η στρατηγικη το 2020. Οπότε και η κρίση έδειξε ποια είναι τα όρια αυτού του εγχειρήματο. Μας πήρε μια δεκαετία να μπορέσουμε να βρούμε κάποιους βασικούς δείκτες και ποια είναι η αρίστη πρακτική όσον αφορά τα συντοξιδοτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τελικά, όσον αφορά το πρόγραμμα διάσωσης στην Ελλάδα, είχαμε μειώσει των συντάξεων κατά 30% μέσα σε μια εβδομάδα. Και επίσης είχαμε άλλου είδους ε, ε, περικοπές της τάξης και σε Ιταλία και Ισπανία. Τι θέλουμε να πούμε δηλαδή, ότι αν έχουμε τέτοιου είδους ε, φωνικό ούτως ε, σύστημα αποφασιστικότητας ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μια τέτοια στρατηγική μακρόπνοη και να μπορούμε για 10 χρόνια να έχουμε τέτοιους στόχους ε, ε, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου στόχου τόσο μακρόπνου. Δεν νομίζω. Ούτε θα βρισκόμαστε στι διαδράσει που βρισκόμαστε σήμερα, θεωρώ εγώ. Οπότε ε, το δημοσιονομικό σύμφωνο και επίση ε, μια νέα συνθήκη όπω λέμε που θα πρέπει να μα οδηγήσει σε νέα διακυβέρνηση. Όλα αυτά αποδεικνύουν στο ότι μέχρι ενό σημείου απέτυχε το σύστημα τη διακυβέρνηση τη Λισαβόνα. Οπότε θα πρέπει τώρα να κινηθούμε σε κάτι άλλο όλο διαφορετικό και θα τα ξαναπούμε όταν έρθει η ώρα να ολοκληρώσουμε, αλλά τώρα δίνω τη σκητάλη στον συνάδελφο. Um, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο Δημήτρης και να σας πω ότι το γεγονός ότι το ευρώ βρίσκεται σε κρίση αυτό είναι ένα εξωγενές σοκ το οποίο μας επέτρεψε να χαράξουμε μεμονωμένες πολιτικής ε, κυρίως ε, σε σχέση με τους στόχους της Λισαβόνας. Εκείνο λοιπόν που θέλω να κάνω τα επόμενα 10 λεπτά είναι να σας μιλήσω για τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της ε, πολιτικής, για τις απειλές ε, και τους κινδύνους που απορρέουν βέβαια και για κάποιες επιτυχίες. Και νομίζω αξίζει ευθύς εξ αρχής να πούμε ε, ότι τα αποτελέσματα δεν δείχνουν μια τόσο ρόδινη εικόνα για την ε, πολιτική, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πριν από την κρίση του ευρώ, η ε, ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ήταν ιδιαίτερα θετική και η ακαδημαϊκοί που ήταν λιγάκι επικριτικοί περιθωριοποιήθηκαν. Αυτό όμως που μοιάζει τώρα να ισχύει είναι το εξής, ότι καθώς ε, προχωράει η όλη υπόθεση του ευρώ και έχει αλλάξει και η συνθήκη της Λισαβόνας, έχει αλλάξει και η, οικονο... η ακαδημαϊκή συζήτηση. Από πλευράς επιτυχιών θα ήθελα να φερθώ σε τρεις. Η μία επιτυχία είναι ε, κατά εν μέρη ο εξευρωπαϊσμός των προβλημάτων. Το άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα η ε, εθνική πολιτική και το τρίτο που θέλω να πω είναι το θέμα της ε, επέκτασης ή της εμβάθυνσης των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο Δημήτρης, αν δούμε λιγάκι τους ε, αρχικούς στόχους, ε, κανένα κράτος μέλος δεν είναι καλός ε, ποιτητής. Όμως ε, βλέπουμε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε και τι άλλο έχει προκαλέσει η συνθήκη της Λισαβόνας. Τι άλλο πέτυχε η συνθήκη της Λισαβόνας σε όλη αυτή την περίοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξε μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση σε διάφορα επίπεδα, ε, μεγαλύτερη έκθεση σε διάφορες πολιτικές, ιστορίες επιτυχίας ε, στα κράτη-μέλη ε, που αναφέρονται σε διάφορες εθνικές πολιτικές και αυτό κατά την άποψή μου προσφέρει μια συγκεκριμένη δομή και παρά την κριτική που ασκείται ε, όπου υπάρχει σταθερή αναφορά έχουμε ότι το, η γνώση είναι πολύ ψηλότερη. Εξαρτάται βέβαια από το κατά πόσον Υπάρχει και μια συγκεκριμένη πεπατημένη στην ε, στρατηγική απασχόληση που αποκολουθείται. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στο εξή. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει αυτό το γνωστικό πλαίσιο, αυτό όμως συνοδεύεται με δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι η εξή. Παρά την ε, τις πολιτικές που ε, χαράσσονται δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτά γίνονται διεθνείς πολιτικές. Ε, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά. Μερικοί μάλιστα λένε ότι τελικά οι Βρυξέλλες είναι που μιλάνε στις Βρυξέλλες, ότι η Λισαβόνα δεν περνάει μέχρι το εθνικό ή το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ένα άλλο ε, θέμα, η άλλη προϋπόθεση αφορά στο εξής, ότι ο εξευρωπαϊσμός είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Αν δει κανείς ε, την στρατηγική της απασχόλησης ε, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια διαδικασία γνωστική μέσα στην απασχόληση και επίσης θα δει κανείς ότι υπάρχει ένα είδος ε, διαφοροποιημένων επιπέδων, ε, διαφορετικά επίπεδα ε, διαφοροποίησης. Αν δούμε λοιπόν χάρη το θέμα των, της υγείας ή των συντάξεων, θα δούμε ότι εκεί δεν υπάρχει πολύ μεγάλος εξευρωπαϊσμός όπως στην απασχόληση και σε κάποιο βαθμό και στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αν δούμε λιγάκι τις, ε, την δύναμη της σύγκρισης. Τώρα ξέρουμε πολύ περισσότερα για το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Έχουμε πολλές περισσότερες ε, στατιστικές και ενημέρωση από αυτά που είχαμε πριν από τη Λισαβόνα. Υπάρχουν ε, συγκρίσιμα στοιχεία. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να γίνει και πού πρέπει να κατευθυντούμε. Τα κράτη-μέλη είναι πολύ πιο ανοιχτά ε, στις ε, διασυνοριακές συγκρίσεις, ε, στο ότι κάποια άλλα κράτη-μέλη μπορεί να είναι περισσότερο επιτυχημένα και παρά λοιπόν τις δυσκολίες που υπάρχουν παραδείγματος χάρη στο θέμα των συντάξεων, του να συμφωνηθούν κοινέ κατευθυντήρες γραμμές. υπάρχει και μία εξοικείωση που αποδείχθηκε ότι είναι πολύ χρήσιμη. Και θα επανέλθω στο θέμα αυτό, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αποδείξει πάντα κάτι χειροπιαστό που να το αποδίδει άμεσα στη Λισαβόνα. Και από πλευράς ε, επέκτασης των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ε, σκεφτούμε λιγάκι την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, το 96 και την διάχυση των επιπτώσεων αυτής της πράξης, των την αισιοδοξία που διεισδύει ε, σε πάρα πολλούς άλλους ε, τομείς. Αυτή είναι η κλασική διάχυση, είναι η ιδανική περίπτωση για να την αποδείξει κανείς. Και αν δούμε λιγάκι τη στατική της Λισαβόνας, πρέπει να διορτιτούμε. Ε, προχωράει η διαδικασία της ολοκλήρωσης, υπάρχει μήπως εμβάθυνση. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν συνέβη οι συντάξεις και ο τομέας της υγείας ε, δεν περιλαμβάνονται στη στρατηγική της ε, Λισαβόνας και μόνο εφόσον κοιτάξει κανείς το κοινωνικό στοιχείο της ε, Λισαβόνας, αυτό πράγματι μπορεί κανείς να το εντοπίσει και πάλι σε θέματα απασχόλησης ε, και θέσεων εργασίας. Όσον αφορά λοιπόν τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, δεν βλέπουμε να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Πάμε τώρα στις ε, αδυναμίες μπορούμε να μιλάμε για ε, γνωστική μετατόπιση, αλλά στην ε, πραγματικότητα η συνθήκη της Λισαβόνας δεν καλύπτει τους ε, στόχους της. Και να μπορούμε να διοικηθούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και υπάρχουν εδώ τρία πράγματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Το ένα είναι ότι η στρατηγική της Λισαβόνας ε, ήταν ένας μετακινούμενος στόχος. Δηλαδή παρά τους ε, σαφείς ε, στόχους και την επαναφορά της συνθήκης Λισαβόνας το 2005 η ε, μετακίνηση των στόχων αποδείχθηκε αρκετά προβληματική. Έχουμε λοιπόν την στρατηγική ε, η οποία οδήγησε στη μετατόπιση του τρόπου με τον οποίο η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την κοινωνική συνοχή. Πώς ε, η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί τελικά στην κοινωνική συνοχή. Έτσι το 2000 η συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει ένα είδο πλατφόρμας για τον ευρωπαϊκό εξυγχρονισμό. Επίσης, η στρατηγική επαναφορά της απασχόλησης και της ανάπτυξης το 2005 αυτό οδήγησε σε να υπάρχει και κάποια μετακίνηση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ίσως λοιπόν είναι απαραίτητο ε, να αναπροσδιορίσουμε τους ε, στόχους και αυτό δημιουργήσε πολύ περισσότερη σύγχυση στα κράτη-μέλη. Έχουμε μια ιδεολογική μετατόπιση η οποία μπορεί να βοήθησε τις κυβερνήσεις το 2005 όμως ε, δεν αναφέρει το τι ακριβώς συμβαίνει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, οι οποίοι άμεσα ενδιαφερόμενοι εν μέρη ευθύνονται και για την εφαρμογή της ε, πολιτικής. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον, αν δει κανεί την αναθεώρηση της ε, Europe 2020 οι στόχοι πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούν πράγματι να υπονομεύσουν την ε, ικανότητα των εθνικών φορέων να προχωρήσουν προς την επίτευξη των στόχων. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι ε, το OMC είναι ε, μια δύναμη μορφή διακυβέρνησης Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν ονοματίζουμε τα κράτη-μέλη αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίμαχο στα, ε, στο Συμβούλιο κυρίως. Και ίσως αυτό να έχει οδηγήσει σε κάποιες επιπτώσεις. Πρόκειται όμως κυρίως για, μια, για πολιτικές επιπτώσεις. Η εικόνα που προκύπτει σε σχέση με την ε, Λισαβόνα είναι ότι έχουμε μια κατάτμιση Και αυτή όλη η διαδικασία ε, του να υπάρχει μια ολοκληρωτική εικόνα για την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι ε, θετική. Και κάτι τελευταίο το οποίο προέκυψε και από την έρευνα είναι το εξής. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ε, μιλάμε για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι ένα από τα θέματα που προέχει είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη θεσμικής ε, καθοδήγησης. Τα κράτη-μέλη είναι σε έλεγχο αυτής της ε, διαδικασίας. Ε, όμως αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν επιθυμεί να εκχωρήσει αρμοδιότητες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να αποδείξουν την κυριαρχία και να ενθαρρύνουν ε, τους ευρωπαϊκούς θυσμούς προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν αυτό το οικοδόμημα, ε, το Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο ε, προσπαθεί να κυριαρχεί σε μια τόσο περίπλοκη ατζέντα. Οι συναντήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ασχολούνται με πιο πιεστικά θέματα. Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση έτσι ώστε να προκύψουν και τα, τα ευκταία αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει και αρκετές αρμοδιότητες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ε, καλύψει αυτό το έλλειμμα που υπάρχει. Και ένα τελευταίο θέμα που νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε εδώ είναι ε, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, που είναι ένας κλειστός θεσμός. Και νομίζω αυτό θέτει σε κίνδυνο και την ε, μέθοδο συντονισμού. Δηλαδή ένα από τα βασικά στοιχεία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας είναι να συμπεριλαμβάνει μία σειρά ε, παικτών ε, και αυτούς να τους προβάλλει προς τα έξω. Όμως η ευθύνη αποδίδεται σε πιο κλειστούς ε, θεσμούς και ε, υπάρχει λοιπόν περιορισμός ε, των ε, δυνατοτήτων να δημιουργούνται συνασπισμοί και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι τελικά το OMC δέχεται αρκετά έντονη κριτική για το ότι δεν είναι τόσο δημοκρατικό ε, όσο θα έπρεπε. Σε γενικές λοιπόν γραμμές νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής ε, συμπεράσματα. Η εικόνα της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλωθεί και ένας από τους ε, παράγοντες που έπαιξαν ρόλο είναι η ανικανότητα των κρατών μελών να επιτύχουν τους στόχους της Λισαβόνας. Αυτή η πόλωση είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, διότι ε, περιορίζει, παραδείγματος χάρη, τα κίνητρα για σύγκληση ανάμεσα στα κρατημέλη. Ε, ε, ε, είναι αυτό πολύ επώδυνο για κάποιους στρατηγική της Λισαβόνας αποδεικνύει ότι η διακυβερνητική συνεργασία έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της και έτσι ε, πρέπει να ζητηθούν νέα εργαλεία και νέα συγκεκριμένα μέτρα για να επιτευχθούν στόχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, εμείς ε, είμαστε αισιόδοξοι και παραμένουμε αισιόδοξοι όσον αφορά την Ευρώπη 2020. Οι πρωτοβουλίες οι εμβληματικέ πρωτοβουλίες είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και επειδή διαιτήθενται όλο και περισσότερο πόροι προς τους στόχους της Ευρώπης 2020 και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Πολλοί από τους στόχοι, στόχους της Ευρώπης 2020 μπορούν να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή πολιτική. Η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά το να συνδυάσει τις πολιτικές με την Ευρώπη 2020. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να επιτύχει όλα αυτά σε μια περίοδο λιτότητας. Είπα Είπαμε λοιπόν ότι ε, η επίτευξη του στόχου, των στόχων της Λισαβόνας ε, θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος και να μην θεωρούμε ότι είναι απλά μια συνταγή για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα τα οποία μας παρουσιάζεται όσο αφορά τα επιστημονικά αποτελέσματα. Προτείνω λοιπόν, επειδή δεν περνάει η ώρα, προτείνω να ε, κάνουμε μόνο ε, μικρές σύντομες ερωτήσεις για να ακούσουμε και τις άλλες δύο μιλήσεις, η ομιλήση, κυρία Γκρέσλε. Οι επιπτώσεις ε, από την χωρίς κονδυλίων δεν πιστεύετε ότι είναι μετρήσιμες. Μπορεί κανείς να μετρήσει τα αποτελέσματα. Άλλος παρακαλώ, θέλει κάποιος άλλος να ερωτήσει κάτι, από ό,τι βλέπουμε όχι. Αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε πώς μετρώνται τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις από την χορήγηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε ήδη προηγουμένως νομίζω ότι το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση ε, προβλημάτων οικονομικής διακυβέρνησης κυρίως δεν αρχούν. Νομίζω ότι ορισμένοι προλαλήσαντες ανέφεραν την ανάγκη με, μεγαλύτερων μεταφορών από χώρε που πηγαίνουν καλύτερα προς εκείνες που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά. Βεβαίως αναγνωρίζεται στο γεγονός ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να πουλήσει εύκολα ε, στο κοινό αυτών των χωρών που θα κάνουν τις μεταφορές. Εκείνο το οποίο είναι πιο σημαντικό πιστεύω από το ποσό των χρημάτων που ξοδεύει η Ευρώπη είναι κατά πόσον είναι αποτελεσματικός ο τρόπος. Και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι ήμοι ε, διακυβερνητικές ανοιχτές μεθόδους ε, συντονισμού δεν απέδωσαν. Συνεπώς ε, δεν έχει σημασία αν ε, ο προπολογισμό της Ευρώπης ξοδεύει ένα Ευρώπη. Αν δεν ξοδευτεί σωστά θα πρέπει να ξαναδούμε τι γίνεται. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να ξοδεύει περισσότερα και με καλύτερο τρόπο. Ο μόνος τρόπος που βλέπω δεν είναι κάτι το πολύ επιστημονικό, αλλά να βρει κάτι ε, με το οποίο θα δεσμεύονται τα κράτη-μέλη. Ένα μεταρρυθμιστικό πακέτο ούτω ώστε να προχωρήσει η Ευρώπη. Ας δούμε κάτι το οποίο αναφέρατε, ότι χρειάζονται μεταφορές από χώρες πλεονασματικέ προ τι άλλε. Έγινε μία συγκρίση με το αμερικανικό μοντέλο. Το αμερικανικό μοντέλο όμως, εκεί δεν γίνονται μεταφορές, αλλά υπάρχουν μετακινήσεις αν θέλετε από τις ευέλικτες αγορές εργασίας από τις μεγάλες λίμνες προς την Καλιφόρνια για παράδειγμα. Τώρα, εάν δούμε την πολιτική συνοχή ήμουν εισηγητής για τα ποσοστά απορρόφησης και είχαμε αυτή τη σκανδαλώδη κατάσταση όπου βλέπουμε ότι οι χώρες δεν απορροφούσαν τα κονδύλια. Για παράδειγμα η Ελλάδα πριν από την κρίση δεν απορροφούσε τα κονδύλια. Η Σικελία, Καλαβρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία αλλά δεν είναι σωστό ότι τα χρήματα δεν μπορούσαν να απορροφηθούν, διότι υπήρχε χρηστή διακυβέρνηση, καλές πρακτικές, όπως στην Εσθονία, στην Πολωνία. Η Πολωνία ξεκίνησε με προβλήματα, κατόπιν να έγιναν μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Συνεπώς δεν είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμπόδισε στη χρήση, την αποτελεσματική χρήση των χρημάτων. Υπάρχει υπευθυνότητα. Ή την ευθύνη την έχουν εκείνοι οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια, συνεπώς την έχουν τα κράτη-μέλη. Και όπως είπατε, εδώ δεν χρειάζονται περισσότερα χρήματα, πολύ σωστά, αλλά καλύτερος τρόπος να δαπανηθούν. Ε, αν δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες, είναι δύσκολο και αν δούμε τις μακροοικονομικές συζητήσεις που γίνονται σε επιστημονικό επίπεδο, έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν υπογραμμίζεται αρκετά. Ε, λοιπόν, παραμένουμε πάντοτε ε, στον παλιό ευρωπαϊκό τρόπο των μηχανισμών μεταφοράς και δεν εστιάζουμε στην πολιτική η οποία έχει ως άξονα την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων ευκαιριών και ούτω καθεξής. Τι πιστεύετε εσείς από αυτού. Ε, θα κάνω τώρα. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Δηλαδή, ε, έχουμε βεβαίως την ανικανότητα των κυβερνησίων και των κρατών μελών να δαπανίσουν ε, χρήματα που τους έχουν ε, διατεθεί. Υπάρχει το θέμα της Λισαβόνας και της Ευρώπης 2020. Αυτές οι δύο διαδικασίες δεν διαχέονται ικανοποιητικά στην κοινωνία των πολιτών και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι λένε, οι Βρυξέλλες μιλάνε στον εαυτό τους. Εάν λοιπόν πραγματικά θέλουμε να πιέσουμε προς κάτι όπως είναι η Ευρώπη 2020, ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν. Πρόκειται για όλους τους ε, ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς ε, που φτιάχνουν μια συγκεκριμένη διαδικασία και όπως σας είπα το βρίσκω ενδιαφέρον που βρίσκομαι εδώ και μιλώ για στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Και γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να επεκτείνουμε την στράτευση για αυτά τα θέματα. Επίσης, όταν σκεπτόμαστε για την κινητικότητα της εργασίας και την ελεύθερη μετακίνηση ατόμων, η γλώσσα στις ΗΠΑ είναι τα αγγλικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε γλωσσικούς φραγμούς. Έτσι λοιπόν ένα πρόβλημα με την κινητικότητα της ε, απασχόλησης σε παρήματος χάρη προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η πλειοψηφία των ε, μεταναστών στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου οδήγησε στο να χάσουν ε, κάποιες δεξιότητες γιατί δεν έχουν την γλωσσική ικανότητα έτσι ώστε να μπορούν να αποδίδουν όπως κάποιοι άλλοι. Εάν λοιπόν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της κινητικότητας θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το θέμα των γλωσσικών δεξιοτήτων και την ποιότητα της γλωσσικής εκπαίδευσης που θα επιτρέψει την κινητικότητα στην ε, απασχόληση. Γιατί μέχρι τώρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος ε, να ρωτήσει κάτι. Από ό,τι βλέπω όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Κόπλαντ. Τα λέμε. Ja, ich komme damit äh, zum dritten Teil der... Έρχομαι λοιπόν στο τρίτο σκέλος του σημερινού απογεύματος και θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθουν εδώ ε, στο βήμα ο κύριος Χένρικ Οτμπό από το ε, ελεγκτικό συνέδριο και ο Δόκτωρ Μάνουελ Μάτες. Ε, τώρα θα εξετάσουμε το θέμα κατά πόσον ήταν επιτυχημένη η στρατηγική που ακολουθήθηκε και θα θέλαμε να έχουμε και μια ποιοτική αξιολόγηση. Θα ήθελα λοιπόν Να καλωσορίσω το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου και εφόσον το επιθυμείτε θα ήθελα και να σας δώσω και το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πια και μέλη τη Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η τελευταία συνεδρίαση τη Επιτροπή σα πριν από τι εκλογέ. Συνεπώ, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ το ελεγκτικό συνέδριο σήμερα και να σα παρουσιάσω μία ανεξάρτητη εικόνα με βάση το έργο που επιτελεί το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, λαμβάνω υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς, γι' αυτό θα σας κάνω μια πολύ σύντομη, συντομότερη ομιλία ό,τι είχα προβλέψει. Βλέποντα τη στρατηγική τη Λισαβόνα, νομίζω ότι ο καλύτερο τρόπο να αξιολογήσει κανεί τα αποτελέσματα είναι να εστιάζεται όχι μόνο σε εκείνα τα οποία δεν επέτυχε η στρατηγική τη Λισαβόνας, αλλά στα διδάγματα που μπορεί κανεί να αποκομίσει. Ποια είναι τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε για να έχουμε καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το πλαίσιο της Αττικής Λισαβόνας και ορισμένα παραδείγματα για την προσαρμογή της. Κατόπιν θα δω τις αξιολογήσεις που έγιναν από την Επιτροπή τις βασικές αδυναμίες ε, της, στην εφαρμογή στρατηγικής, όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα στο ελληνικό συνέδριο, και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα μελλοντικά προγράμματα. Η γραπτή μου ομιλία αναφέρει πολλά παραδείγματα ε, των ελέγχων που έχει κάνει ε, το ηλεκτρικό συνέδριο, αλλά δεν μπορώ τώρα στην προφορική μου παρουσίαση να σας τα δώσω όλα. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η στατική της αφορά όλη την Ένωση. Και βεβαίω τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής μπορεί, δεν μπορεί να, επηρεάσει την υλοποίηση των στόχων στρατηγική. Η στρατηγική της Αγώνα είχε ως σκοπό να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την πιο δυναμική οικονομία στον κόσμο με βάση τη γνώση, ικανή ε, μιας βιώσιμη με, με περισσότερες δουλειές και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον μέχρι το 2010. Αυτοί οι ευρωπαϊκοί στόχοι, όπως είπαν πολλοί ομιλητές σήμερα, εκπροσωπούν μια προσέγγιση η ενιαία προσέγγιση δεν ε, λάμβανε υπόψη τις ε, αδυναμίες και τα δυνατά σημεία των κρατών μελών και τώρα εκ των υστέρων βλέπουμε ότι αυτή η προσέγγιση καθορισμού στόχων μπορεί να συνέβαλε ε, στην έλλειψη κυριότητας όπως τα λέγαμε σε δίκη της Αβώνας. Η πρώτη φάση της στρατηγικής εστιαζόταν στην ήθελε να μεταφράσει ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε μέσα πολιτικής. Αυτό γινόταν με προσανατολισμούς πολιτικής, όπως στην κοινωνία της πληροφόρησης, στην έρευνα και ανάπτυξη. Με βάση την ενδιάμεση αξιολόγηση που έγινε τον Νοέμβριο του 2004, η Επιτροπή κατέληξε ότι τα αποτελέσματα μέχρι τότε ήταν απογοητευτικά και ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν κατόρθωσε να δώσει τα στοιχεία που αναμένονταν όσον αφορά την παραγωγικότητα και την απασχόληση. Μετά από αυτή την ενδιάμεση αξιολόγηση η Επιτροπή αποφάσισε να εστιάσει την προσοχή της στην αύξηση των θέσεων εργασίας και ξεκίνησε με τέσσερις τομείς προτεραιότητας. Έρευνα και καινοτομία, επένδυση στους ανθρώπους, μεγαλύτερη επιχειρησιακή ικανότητα και ενέργεια και κλιματικές αλλαγές. Ενώ το 2007 ήταν θετικό όσον αφορά την ανάπτυξη και την καθαρή απασχόληση, άρχισε, ξέσπασε η κρίση και, και δημιουργήθηκαν άλλε προτεραιότητες. Η μεγαλύτερη προτεραιότητα ήταν να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου πολίτες από τις φοβερέ επιπτώσεις της οικονομική κρίσης. Η πρόσβαση των ιδιωτικών επιχειρήσεων ε, σε χρηματοδότηση ήταν προτεραιότητα. Αυτό, αυτή ήταν προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν απασχολήσεις στον ιδιωτικό τομέα η έρευνα και η καινοτομία και επίσης υποδομές στην ενέργεια, σε επενδύσεις, όλα αυτά αυξήθηκαν. Θα ήθελα να σα δώσω ορισμένα παραδείγματα με βάση τους ελέγχους που έχουμε διενεργήσει. Το 2012 το συνέδριο ε, δημοσίευσε μια έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγχρωματοδοτούμενο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης. Δυστυχώς υπήρχαν πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω ε, του ρυθμιστικού πλαισίου που δεν ήταν ανεπαρκές, της ανεπαρκούς ανάλυσης των αναγκών και ατελούς παρακολούθησης του συστήματος αξιολόγησης. Επίσης, έπρεπε να γίνουν επενδύσεις, ενέργεια, σε ενεργειακή απόδοση και καταλήξαμε ότι οι προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν σωστή ενεργειακή απόδοση δεν είχαν εξασφαλιστεί. Δεν υπήρχαν σωστές αξιολογήσεις για να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας και δεν είχαν ενσωματωθεί στα εθνικά προγράμματα ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη, πιστεύω ότι μπορώ ασφαλώς να καταλήξω, όπως έκανε η Επιτροπή το 2010, ότι η Στατική Λισαβόνας δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τους στόχους απασχόλησης και ανάπτυξης. Συλλογικά τα κράτη-μέλη δεν κατόρθωσαν να κλείσουν αυτό το χάσμα παραγωγικότητας που είχαν με τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Οι συνολικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στα κράτη-μέλη και τα στοιχεία απασχόλησης σημείωσαν βελτίωση πριν από την οικονομική κρίση του 2008. Ενώ κανένας μεμονωμένος έλεγχο δεν θα μπορούσε να εκτιμήσει τις συλλογικές επιπτώσεις της στρατηγικής Λισαβόνας, το λεκτικό συνέδριο προσπάθησε να δώσει τα στοιχεία που μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη. Ενώ οι έλεγχοι του ελεκτικού συνεδρίου σημείωσαν ορισμένα ωφέλη για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες, Αυτά τα ωφέλη θα ήταν μεγαλύτερα ε, και με χαμηλότερο κόστος εάν ήταν καλύτερα στοχευμένη και προγραμματισμένη η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είδαμε ότι σε ορισμένου τομείς τα αποτελέσματα δεν μπορούν να μετρηθούν και να τεκμηριωθούν επειδή δεν υπάρχουν στα στοιχεία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα διότι δεν επιτρέπει τον έγκυρο προσδιορισμό της κακής απόδοσης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Επίσης, δεν μπορούμε σωστά να προβλέψουμε τα μελλοντικά προγράμματα και περιορίζει ε, την ε, ικανότητα της Επιτροπής να επιβάλλει φορολογικά μέτρα. Έχουμε ένα νέο κεφάλαιο τώρα που αφορά την απόδοση και τους πόρους που θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση την έκθεση επίδοσης, κάθε χρόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με διαχείριση. Ένα από τα θέματα είναι η προστιθέμενη αξία, που μερικές φορές υπήρξε ένα δύσκολο στοιχείο όταν προγραμματίζει τους ελέγχους στο Ελληνικό Συνέδριο. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο προκύπτει σε πολλούς ελέγχους αναγνωρίστηκε και στην ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής Λισαβόνας είναι το πρόβλημα να έχει κανείς αποτελέσματα σε τομείς όπου δεν υπάρχουν επαρκείς στόχοι ε, και δείκτες για τα λειτουργικά προγράμματα. Αυτές είναι προϋποθέσεις για να παρακολουθεί κανείς ε, την εξέλιξη των προγραμμάτων. Ο νομοθέτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν σαφείς στόχοι πολιτικής. Διότι αν δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι πολιτικής, τότε θα δαπανώνται χρήματα άσκοπα, θα υπάρχουν ε, αντικρουόμενες πρωτοβουλίες. Αλλά όταν υπάρχουν σαφείς στόχοι πολιτικής, στους κανονισμούς, τα πράγματα είναι ευκολότερα, δεν αρκούν. Η Επιτροπή και τα κρατη πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον καθορισμό εστιασμένων στόχων, καθώς και στον τρόπο περιορισμού των κινδύνων όταν οι στόχοι δεν υλοποιούνται. Ορισμένοι έλεγχοι που έχουμε επιτελέσει ε, εστιάστηκαν σε δείκτες, αλλά δεν εφαρμόστηκαν με συνέπεια στα τελευταία προγράμματα. Σε, ορισμένους, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι ώστε να, ε, να, μπορούμε να, να μετρούμε τα αποτελέσματα ετησίως. η μέτρηση και αξιολόγηση της πραγματοποίησης των στόχων καθίσταται δυνατή μόνον εάν υπάρχει ένα παρκές σύστημα στο ξεκίνημα του προγράμματος, ικανό να δώσει στοιχεία αξιόπιστα. Με την έναρξη της νέας προγραμματικής περίοδου, το Λεδικό Συνέδριο υπογραμμίζει την ανάγκη διαχείρισης των επιδόσεων και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νομικοί περιορισμοί και οι πρακτικοί περιορισμοί δεν εμποδίζουν την παροχή αξιόπιστων στοιχείων όσον αφορά τα προγράμματα και τη διαχείριση αυτών. Η Επιτροπή επίσης πρέπει να δει πώ θα εξασφαλίζει ότι οι κατάλληλε πληροφορίες θα παρέχονται την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για την έκθεση Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης. Αυτή η πολύ σημαντική έκθεση, ετήσια, αυτή τη στιγμή δεν εκπληρεί ε, τις προϋποθέσεις. Συνεπώς, το Λιτικό Συνέδριο εξηγεί πώς μπορεί η έκθεση να δώσει πιο αξιόπιστες πληροφορίες και όσον αφορά τα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία εξασφάλισης καλύτερων, ε, παροχής καλύτερων και έγκαιρων στοιχείων στις γενικές διευθύνσεις και να λαμβάνει υπόψη τους στόχους τους παραλήπτες και τις διασυνδέσεις μεταξύ ε, των ε, μηχανισμών ελέγχου. Συνεπώς, θεωρώ θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή το 2013 δεσμεύτηκε να παρουσιάσει φέτος, το 2014, ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση απόδοσης ε, και την υποβολή εκθέσεων. Το ελληνικό συνέδριο θα εξακολουθεί να παρακολουθεί και να δίνει αφορά σχετικά με την επιτυχία της Επιτροπής. Τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση θα ήθελα να υπογραμμίσω τα βασικά στοιχεία. Δεδομένου ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει στην αξιολόγηση τη στρατηγικής τη Λισαβόνας 2010 τους στόχους, ότι οι στόχοι ανάπτυξης και απασχόλησης δεν υλοποιήθηκαν από τα κράτη-μέλη, πρέπει να υπογραμμίσουμε τους λόγους καθώς αναφέρουν οι έλεγχοι του Ελληνικού Συνεδρίου, τα προγράμματα δαπανών δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους και στους δείκτες. Δεν υπήρχε σωστό σχεδιασμός και προγραμματισμός και δεν υπήρχε ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης των αποδόσεων. Αυτές οι αδυναμίες περιορίστηκαν σημαντικά θα έπρεπε να πούμε με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ότι η διαχείριση απόδοσης και της υποβολής ε, αναφορών εξελίσσεται. Αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη η Επιτροπή. Χρειάζεται την υποστήριξη του νομοθέτη και τη δέσμευση των κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή πρέπει να εξακολουθεί να υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη την υποχρέωσή τους να χρησιμοποιούν τα ε, ευρωπαϊκά κεφάλαια σύμφωνα με ένα σωστό πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης. Θα πρέπει οι δαπάνες να προορίζονται ε, στα projects τα οποία αποδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η πραγματική δοκιμή θα είναι κατά πόσον η Επιτροπή θα κατορθώσει στη νέα προγραμματική περίοδο να εξασφαλίσει εστιασμένους στόχους με αντίστοιχους δείκτες ούτως ώστε να παρακολουθεί και να μπορεί να μετρήσει τις αποδόσεις και σε ποιο βαθμό είναι ικανή να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020. Αυτοί οι στόχοι, όπως και εκείνοι του 2000 για τη στρατηγική της Αβώνας, θα πρέπει να μεταφράζονται σε συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες στα κράτη-μέλη, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει μια εστιασμένη εφαρμογή, ούτως ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση. Η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα κράτη-μέλη. Ένα σημαντικό ρόλο συνεπώ τη Επιτροπή είναι να συντονίσει την εφαρμογή και να έχει ένα υγιέ σύστημα οικονομική διαχείριση. Το ελεκτικό συνέδριο για τους στόχους 2013-2017 περιλαμβάνει τη μεγιστοποίηση της συμβολής της για τη βελτίωση της λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ελληνικό συνέδριο θα εξακολουθεί να παρέχει στους ενδιαφερόμενους εγκαίρως εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει τα κράτη-μέλη. Επίση, θα εξακολουθούμε να αναφέρουμε τις επιδόσεις και να έχουμε μια ολιστική εικόνα τόσο όσον αφορά τη συμμόρφωση και την επίδοση των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.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 ε, αυτές τις ε, συζητήσεις. Ε, συζητήσαμε πάρα πολύ για την επιτυχία την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας και εγώ θα προσπαθήσω να περιορίσω αυτά που λέξαν και κατά την άποψή μου είναι περιτά. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να συστηθώ. Εγώ ασχολούμαι στο Πανεπιστήμιο της Νιρεμβέργης με τη στρατηγική της Λισαβόνας και δεν ασχολούμαι τόσο με εμπειρικές έρευνες για το κατά πόσον έχουν επιτύχει τα μέτρα, αλλά ασχολούμαι περισσότερο με το περιεχόμενο της στρατηγικής. Πρόκειται για ένα θέμα το επί το οποίο σήμερα δεν έχουμε εμβαθύνει. Και γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι αυτά που σας πω είναι μια χρήσιμη προστίκη. Στην έρευνά μου την προσοχή μου στο κατά πόσον το οικονομικοπολιτικό πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί μια προϋπόθεση για να υπάρχει μια ικανοποιητική εξέλιξη στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι στόχοι της στρατηγικής, δηλαδή η διασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακούσαμε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έχει ένα ευρύτατο πλαίσιο και η βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης είναι ένα μόνο κομμάτι αυτής. Βεβαίως ε, είναι σκόπιμο να προβάλλει κανείς ε, όλα τα θέματα, κυρίως ε, κατά τη διαμόρφωση στρατηγικής του, που έλαβε χώρα αυτό το 2005. Θέλησα να εξετάσω το κατά πόσον η στρατηγική ενδείκνυται πράγματι για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει κανείς εδώ να αντιρωτηθεί ποιοι είναι ε, οι βασικοί παράγοντες, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις ε, πάνω στις οποίες βασίζεται η στρατηγική. Και αν μπει κανείς λιγάκι την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο διαπιστώνει ότι τα βασικά στοιχεία ή το βασικότερο στοιχείο είναι η έλλειψη ευέλικτων ισοτιμιών. Και αυτό προκλήθηκε από την νομισματική ένωση. Βεβαίω και υπάρχουν χώρε που δεν έχουν ε, υιοθετήσει ακόμα το ευρώ, αλλά ο στόχο είναι το ευρώ να γίνει τελικά ε, το νόμισμα του συνόλου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και προκλήσεις που αφορούν στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δει λοιπόν κανείς ε, τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο από μια εξωτερική διάσταση θα καταλήξει στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη ε, με όλο και περισσότερο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται αντιμέτωπες με ανταγωνιστές οι οποίοι παράγουν σε άλλο οικονομικό χώρο και έχουν ε, προϋποθέσεις παραγωγής ε, που αποκλίνουν από τις συνδυσμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι βέβαια οι ε, παράγοντες παραγωγής, οι τιμές που συμβάλλουν καθοριστικά στο ποιοι τομείς μπορούν να επιμερίσουν καλύτερα στον οικονομικό χώρο. Υπάρχουν λοιπόν δύο προκλήσεις. Υπάρχει ο μηχανισμός των ευέλικτων ισοτιμιών. Αυτός ο μηχανισμός ε, δεν υφίσταται πια και η δεύτερη πρόκληση είναι να βρεθούν απαντήσεις ε, στον όλο και μεγαλύτερο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ας δούμε λοιπόν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις. Απαντήσεις υπάρχουν στην οικονομική βιβλιογραφία. Αριστερά βλέπετε και πολλοί θα γνωρίζετε ότι η θεωρία αναφέρει τους βέλτιστους ε, νομισματικούς ε, χώρους. Το τι δηλαδή πρέπει να καλύπτεται ως κριτήριο για να έχουμε το βέλτιστο νομισματικό χώρο. Και όσο καλύτερα καλύπτουν τα κριτήρια αυτά, τόσο καλύτερα μπορεί κανείς και να αποφύγει τις ανομαλίες, τα σοκ, τις διαρθρωτικές διαφοροποιήσεις, αλλά και τις διαφορές στον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μόνο ένας νομισματικός χώρος που έχει εναλλακτικές λύσεις προσαρμογής, μόνο αυτός μπορεί μπορεί να αντιμετωπίσει τα οικονομικά σοκ. Και θα ήθελα να αναφέρω και κάποια παραδείγματα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στη συζήτηση που κάναμε ε, ελέγχθησαν ορισμένα πράγματα, παραδείγματο χάρη η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, που κατ' ουσίαν αν θέλετε είναι ο μηχανισμός ε, προσαρμογής, ε, ο οποίος ε, είναι και ο σημαντικότερος διότι με αυτή τη θεωρία ε, δημιουργήθηκε ακριβώς αυτός ο μηχανισμός. Η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει στο να μην υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού ένα νομισματικό χώρο. Δεύτερος μηχανισμός προσαρμογής, ευελιξία των μισθών. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, οι μισθοί έχουν πέσει σημαντικά ή πιέστηκαν αν θέλετε σημαντικά λόγω της λήψης πολιτικών μέτρων. Η Ελλάδα βέβαια αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υποτιμήσει το νομίσμα της. Και ακριβώς αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, μείωση των μισθών ενδέχεται η Ελλάδα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, αλλά αυτό που είναι καθοριστική σημασία είναι οι συσχετισμοί ε, μέσα στον ε, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Χώρο. Δηλαδή η αναλογικότητα και η σχέση των ελληνικών με τους γερμανικούς και τους γαλλικούς μισθούς. και σε τελική ανάλυση οι μισθολογικές ε, εξελίξεις ε, όσο και αν πλήττουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ε, δικά για την δουλειά της Ελλάδας πρέπει να σου πω ότι η πτώση των μισθών θα βοηθήσουν, θα βοηθήσει στο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι μηχανισμοί προσαρμογής. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ένα παράγοντα, παρότι έχει περάσει η ώρα, ε, με συντονισμένη οικονομική πολιτική ε, είναι δυνατόν ε, να προλάβει κανείς κάποιες εξελίξεις και επίσης μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει και αποκλίσεις. Συνοπτικά θα έλεγα το εξής, ότι όσο καλύτερα καλύπτει ένας νομισματικός χώρος όλα αυτά, την προσαρμογή αν θέλετε, τόσο πιο σταθερός είναι και τόσο ε, καλύτερες είναι και οι προϋποθέσεις των επενδύσεων. Δεξιά, εκεί που γίνεται λόγος για τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και αυτό αναφέρθηκε σήμερα, της ε, σχετικής ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή πρόκειται για το εξής. Η οικονομική βιβλιογραφία μας αναφέρει ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να οδηγήσει στην διεθνή εξειδικευσή και κυρίως σε αυτούς τους τομείς όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το ερώτημα που έθεσα είναι το εξής. Κατά πόσον τα κριτήρια αυτά καλύπτονται από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Και αν δει κανείς τα κριτήρια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο της στρατηγικής της Λισαβόνας ανταποκρίνεται μια χαρά σε αυτές τις απαιτήσει. Ε, στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αυτό που βλέπετε αριστερά, και επίση και να βρεθεί μια απάντηση στο διεθνή ανταγωνισμό με νέες τεχνολογίες, ε, κυρίως ε, εφόσον κανείς ε, θεωρεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ε, ελπιδοφόροι τομείς του μέλλοντος που πρόκειται βεβαίω για ε, τομείς έντασης κεφαλαίου. Και θα αναφέρω εδώ κάποια παραδείγματα. Μιλήσαμε για τη μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού. Νομίζω όμως ότι με τη μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, ένα εξορθολογισμό της ε, πολιτικής, ε, την παρεμπόδιση των αντιφάσεων και επίσης η μέθοδος του ανοιχτού συντονισμού προσφέρει τη δυνατότητα να συμβάλλει κανείς με διαρθρωτικές διαφορές και σε τελική ανάλυση η μέθοδος αυτή ενισχύει την συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να φερθώ και σε ένα άλλο, σε θέμα, στην οδηγία περί παροχής υπηρεσιών η οποία οδηγία αυτή εισήχθη κατά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Και αυτή η οδηγία ενδείκνυται έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του οικονομικού και νομισματικού χώρου, επειδή προάγει την κινητικότητα των εργαζομένων. Όχι βέβαια μακροπρόθεσμα, ε, διότι η παροχή υπηρεσιών είναι αν θέλετε κάτι το πρόσκαιρο, όμως ε, γενικά ε, προάγεται η κινητικότητα των εργαζομένων. Επίσης και τη ροή κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε με την ε, Λισαβόνα, τη συνθήκη της Λισαβόνας, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ροή κεφαλαίων στην Ευρώπη. Επίσης ενδείκνύται και οι οικονομικές ε, μεταφορές ε, έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα όπου σε εκείνες τις χώρες όπου δεν υπάρχει ικανοποιητική ανταγωνιστικότητα, ειδικά στις χώρες αυτές γίνονται επενδύσεις Δεξιά λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια κοινωνία της ενημέρωσης, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου. Όλα αυτά τα μέτρα ενδείκνυνται έτσι ώστε να επενδυθούν κονδύλια, κυρίως ιδιωτικά κονδύλια, σε τομείς οι οποίοι ενδείκνυνται ιδιαίτερα ε, για να υπάρχει επιμερία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική της Λισαβόνας ακολουθεί σαφώς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως η εικόνα αυτή ε, αμαυρώνεται κατά τη από μια ημιτελή εφαρμογή των μέτρων. Μιλήσαμε παραδείγματο χάρη για την οδηγία παροχή υπηρεσιών. Αυτή λαμβάνεται ως κριτήριο για τι προκλήσει που προανέφερα. Και βεβαίω ε, αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, το να διευθυνθούμε το τι θα γινόταν αν εφαρμοζόταν η αρχική μορφή της οδηγίας περί παροχής υπηρεσιών. Ε, διότι ε, με τον τρόπο αυτό ενδεχομένω να είχε απλουστευτεί κατά πολύ η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Ε, το σχέδιο που τελικά εγκρίθηκε δεν επιφέρει την απελευθέρωση και την ευελιξία ε, που ε, αυτό έχει ως στόχο η πρόταση της Επιτροπής. Θα αναφερθώ τώρα στους ε, στόχους, κυρίως ε, στους στόχους που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την αηφορία των δημοσιονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Εδώ υπάρχει μια αντίθετη πολιτική το σύμφωνο της ε, σταθερότητας ε, δεν ενισχύθηκε αλλά αποδυναμώθηκε κατά τη διάρκεια της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Και θα αναφέρω και άλλο ένα παράδειγμα και με αυτό θα κλείσω στο κοινοτικό δίπλωμα ευρεστεχνίας, το οποίο αναφέρεται ως ένα πακέτο για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Ε, τέλος, καταλήγω στο εξής, ότι από πλευράς περιεχομένου η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν μια στρατηγική η οποία αναγνώρισε τις σημαντικές προκλήσεις, όμως δυστυχώς δεν έγινε η σωστή εφαρμογή των μέτρων. Υπάρχει η μέθοδος του ανοιχτού συντονισμού. Η μέθοδος όμως αυτή δεν είναι κοινοτική μέθοδος και δεν θα πρέπει να γύρει κανείς ε, τον ισχυρισμό ότι είναι κοινωτική μέθοδος. Πρόκειται για ένα ε, συντονισμό, συντονιστικό μέσο εθνικών πολιτικών. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το εργαλείο έχει και συγκεκριμένα όρια. Και να πω μόνο ότι όπως και η δημοσιονομική πολιτική δεν κατόρθωσε να επηρεάσει σημαντικά την πολιτική των ε, κρατών μελών. Στη δημοσιονομική πολιτική υπήρχε ένα μέτρο κυρώσεων ε, που όμως ε, δεν υπήρξε τελικά στο συντονισμό. Και γι' αυτό η μέθοδος του ανοιχτού συντονισμού αυτή δεν πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν καταλήγω στο ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει εντοπίσει τις σημαντικότερες προκλήσεις, αλλά τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών η στρατηγική αυτή υπολείπεται των στόχων. Και σε τελική ανάλυση, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ε, δεν θα πρέπει να επιμένουμε τόσο πολύ στην Ευρώπη του 2020. Η στρατηγική αυτή βασίζεται κυρίως στην στατική της Λισαβόνας με τις θετικές και τις αρνητικές της πλευρές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Δόκτωρ Μάρτες και κύριε Ότμπο. Και τώρα, ε, αν θέλετε, μπορούν να ξεκινήσουν τα σχόλια. Η κυρία Κρέσλε, καταρχήν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Βλέπουμε λοιπόν ε, ότι υπάρχει κάποια μηχανία ακόμα και στους εμπειρογνώμονες της οικονομίας. Ε, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι ήρθατε. Ε, είπατε ότι να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία και ρωτώ τι πρέπει να κάνουμε καλύτερο στην πολιτική του 2020. Είναι μια ερώτηση και προς τους δύο. Ο κύριος Μούλντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ έχω μια ερώτηση για τον κύριο Όλμπο, αλλά και σχέση με τον κύριο Μάτε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ε, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και συμφωνώ με όσα είπαν να είχαμε κάποιο είδου ε, δείκτε και κριτήρια. Για να μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ κάθε φορά ποιο είναι το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει. Ε, άπαξ βέβαια και το οικονομικό περιβάλλον και η συγκυρία αλλάζουν τόσο γρήγορα, τόσο ώστε το ΑΕΠ ας πούμε της Ελλάδας έχουν επί 20% και της Ιταλίας έπρεπε κατά 10% μα πώς είναι δυνατόν κανείς ποτέ να μπορέσει να υιοθετήσει κάποιου είδους παραμέτρους ε, αξιοπίστους ε, αξιόπιστες τέλος πάντων τόσο να μπορέσει να περιχαραγώσει το πρόβλημα ούτως ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε έτσι κάποιο ε, πρόγραμμα όταν δεν μπορεί να ξέρει κανένα ακριβώ ποια θα είναι η απόδοση του εγχείρηματο κάθε φορά. Ο επόμενο, κύριε Κρίστο. Σας ευχαριστώ λέει κύριε Γκρέσλε. Υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα, το οποίο το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα δύο χρόνια. Κάποια πράγματα πρέπει να καταρτήσουμε. την τάσκο στην Ελλάδα, έχει 180 διαφορετικά προγράμματα, σχέδια. Επίση να δούμε τι έγινε στην Τσεχία πριν από 15 μέρε. Αυτά τα προγράμματα και σχέδια θα πρέπει να εκτελεστούν μέχρι το τέλος. Οπότε θα πρέπει να υιοθετηθεί τέτοια νομοθεσία που να μπορέσει να μην καταλήξει σε κάποια πολιτική αντιπαραγωγική. Τα κρατημέλη όπως είναι σήμερα η συγκύρια δεν μπορούν να έχουν κάποια προοπτική. Άρα τι θα γίνει με όλα αυτά τα προγράμματα και σχέδια τα οποία δεν θα ξεκινήσουν υπό τις καλύτερες συνθήκες. Δώστε κάποια σύντομη απάντηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις κυρία Γκρέσλε και κύριε Μίλτερ, λέει ο κύριος Όντμπο. Πρώτα απ' να δούμε ε, στο ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση κοινοτική μόνο όταν έχουν προσθέμενη αξία. Γιατί σήμερα υπάρχει δυσκολία να μπορέσουμε να ορίσουμε πότε συντρέχουν ε, αυτές οι προϋποθέσεις. γιατί γίνονται δαπάνες και από τους πολύ πιο σημαντικούς ε, από όγκου εθνικούς προπολογισμούς. Θα πρέπει να αναγνωριστεί το ότι είναι σημαντική η συμμόρφωση. Αλλά απομακρυνόμαστε με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό από αυτήν την ε, αντίληψη. Όσον αφορά τη μεταφορά κονδυλίων, την απορρόφηση από τους στόχους γιατί η Ένωση θέλει να υπάρχουν επιπτώσεις, αποτελέσματα από την χρηματοδότηση. Νομίζω ότι μέχρι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι δαπάνες έχουν γίνει με τον επιθυμητό τρόπο. Άρα θα πρέπει να κάνουμε το δύσκολο το να δούμε ποια κριτήρια θα υιοθετήσουμε. Κύριε Μάτες, λέει ο Πρόεδρος, έχετε εσείς το λόγο για να απαντήσετε. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη στρατηγική 2020 επί τη βάση της ανάλυσης που σας εξέθεσα. Νομίζω ότι η στρατηγική της Λισαβόνας σχεδιάστηκε σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε τι προκλήσεις έχουν αντιμετωπιστεί. θα διαπιστώσετε τότε ότι η στρατηγική αυτή δεν έχει λάθος κατεύθυνση. Και όπως και οι προλαλήσαντες, και εγώ θεωρώ, ότι το πρόβλημα είναι η μη ορθή εκτέλεση της στρατηγικής. Άρα εδώ θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πώς θα πρέπει να αλλάξουμε διάφορε πολιτικές, μην έχουμε μόνο ε, νομοθετήματα μη υποχρεωτικά. Επίσης, πολλά θα εξαρτούν από το πόσο αποφασισμένα είναι τα κράτη-μέλη, που δεν είναι αποφασισμένα τη σήμερα ημέρα. γι' αυτό και νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, η συγκήτρια τώρα θα πρέπει να προβεί σε εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Κυρία Γκρέσλε, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για να δούμε τι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει αν δεν υπήρχε η κρίση. Απασχόληση, ανάπτυξη. Ήταν πάρα πολύ πλήρες οι παρεμβάσεις των ε, εισηγητών. Τι θα μπορούσε να μην έχει γίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τροφή προσκέψη οικονομικές πολιτικές, σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνα, σε σχέση με την καινοτομία, τι έγινε σε κάθε κράτος μέλος. Σε κάποια κράτη-μέλη. Οι θέσει απασχόλησης ε, είναι σημαντικές ε, αλλά είναι σημαντικές κυρίως για τον ερευνητικό τομέα. Εκεί καταβλήθηκε η προσπάθεια παντού να υπάρξει πνευματική υπεραξία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε, δηλαδή στις συγκεκριμένες συνέπειες αυτής της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είδαμε ότι τα κονδύλια μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εφόσον υπάρχει επιτυχία. Δηλαδή η στρατηγική της Λισαβόνας ε, θα πρέπει να είναι πολύ πιο επιτυχημένη και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 να μην η στρατηγική αυτή να μην έχει το ίδιο τέλος. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε τελικά να επενδύσουμε στην καινοτομία για να ε, επιδιώξουμε τους ε, στόχους με μεγαλύτερη συνέπεια. Με μεγαλύτερη συνέπεια από ό,τι το κάναμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι εξετάσαμε σήμερα το θέμα αυτό. Υπάρχουν ε, κρατημέλη τα οποία λειτουργούν μόνο μετά από πίεση ε, και πολλοί λένε ότι όλοι μας θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι ε, κυρίως στο ερώτημα του τι θέλουμε να επιτύχουμε. Ο ανοιχτός ε, συντονισμός είναι αυτός που είναι και εγώ έλαβα υπόψη μου ότι το πλεονέκτημα του ανοιχτού συντονισμού είναι ότι προκύπτουν συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ασκηθεί πίεση. Έτσι βλέπαμε εμεί πάντα την αξία του ανοιχτού συντονισμού. Ε, και βεβαίως και το γεγονός ότι ο ανοιχτός συντονισμός μπορεί να γίνει πολύ πιο ουσιαστικός. Ε, η έλλειψη ιδεών συμβαδίζει με την έλλειψη κονδυλίων και τίθεται το ερώτημα τι θα κάνουμε με τους, με τα, με τους τομείς εκείνους όπου δεν υπάρχει υποδομή. Ε, και γι' αυτό ε, δημιουργείται και το θέμα των ιδιαίτερων οικονομικών ζωνών. Ε, νομίζω λοιπόν ότι στο νέο κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ρωτήσουμε κατά πόσον ε, σε κάποιες περιοχές θα πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω. Νομίζω ο Επίτροπος κ. Λεβαντόφσκι είπε ότι η συγκέντρωση ε, σε κάποιες συγκεκριμένες δομές σημαίνει ότι Θα πρέπει οι επενδύσεις ε, να επικρατούν και να γίνεται επένδυση κυρίως ε, στην έρευνα ε, και όχι τόσο στις υποδομές. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι όλοι μας παρουσιάσετε πάρα πολύ καλές ιδέες, τις οποίες εμείς οπωσδήποτε θα τις ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τη γραμματεία που προσπάθησε να σας βρει ε, γιατί θέλαμε να κάνουμε ανάλυση πόλεων και χωρών και τελικά ε, δεν κατορθώσαμε ε, να μας βρούμε αυτούς όλους να θα ενημερώσουν για διαφορα κρατημέλη. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τη Γραμματεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Γκρέσλε και θα ήθελα ως πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμών να δράξω την ευκαιρία γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η τελευταία μας συνεδρίαση κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας του ε, Κοινοβουλίου. Να ευχαριστώ καταρχήν τους ομιλητές του σημερινού απογεύματος. Νομίζω ότι ε, ήταν ιδιαίτερα θετικό το ότι ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας με την αξιολόγηση της ε, στρατηγικής της ε, Λισαβόνας. Γιατί το ότι το θέμα αυτό δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από ό,τι προσφέρει απαντήσει, αυτό είναι αυτονόητο. Και τίθεται το ερώτημα του πώς θα ε, αναπτύσσονται τα κράτη-μέλη αν δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τίθεται το ερώτημα γιατί ορισμένα κράτη με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα από άλλα. Και τίθεται και το ερώτημα για εκείνα τα κράτη τα οποία είναι μέλη της Ευρωζώνης κατά πόσον Πράγματι, τα κράτη αυτά ε, εξελίχθηκαν χειρότερα από άλλα που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης, γιατί υπάρχει πράγμα το εξής ε, περίεργο, ότι κάποια κράτη έχουν το ευρώ και αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά και άλλα που δεν έχουν το ευρώ και αυτά έχουν κρίση. Που σημαίνει ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε για το κατά πόσον το νόμισμα είναι η ειδοποιώ διαφορά ή όχι. Μήπω τα προβλήματα έρχονται περισσότερο από την πραγματική οικονομία. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά κύριο λόγο το δικό μα το καθήκον. Το δικό μα το καθήκον είναι να ελέγχουμε πού ακριβώ διοχετεύονται τα κονδύλια. Και μας εντόθησαν ε, διάφορες συμβουλές και προτάσεις που νομίζω ότι θα αποτελέσουν μια πολύ καλή βάση για τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι θα συνεχίσουν τις εργασίες τους στην Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών. Θα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εκείνους ε, με τους οποίους ε, συνεργαστήκαμε στην Επιτροπή μας και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε όλους μας σε και κατηδίαν ε, συζητήσεις να ανταλλάξουμε απόψεις ε, ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής, εκ μέρους των μελών της Επιτροπής. Ευχαριστώ όλους για την αγαστή συνεργασία, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της Επιτροπής, τα, τους οργανισμούς. Κυρίως ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο. Σήμερα έχουμε παρόντα και μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Ε, ευχαριστώ βεβαίως ε, και τα μέλη της ε, γραμματείας. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς, τα μέλη των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών συνέβαλε καθοριστικά στον δημοκρατικό έλεγχο. Αν δούμε λιγάκι το τι έγινε μετά από πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λήφθησαν δηλαδή περισσότερα διορθωτικά μέτρα, ε, νομίζω ότι καθίσατε σαφές ότι συμβάλλουμε στα κρατημέλη, στην ε, βελτίωση κατάσταση των κρατών μελών και νομίζω οι πολίτες ε, θέλουν να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα χρήματά τους. οποτεδήποτε κάνουμε επιτόπιες επισκέψεις, είναι απαραίτητο να καθιστούμε σαφές τι γίνεται με τα χρήματα των φορολογουμένων. Και τελειώνοντας θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω και αναφέροντας ένα ιστορικό παράδειγμα. Μερικές φορές με ρωτούν κατά πόσον θα καταφέρουμε ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε αισιόδοξο μέλλον. Στη γενέτειρά μου, που είναι και η γενέτειρα της κυρίας Κρέσλε, συζητάμε το κατά πόσον είναι καλό μια συγκεκριμένη περιοχή να χρηματοδοτεί μια άλλη όπως είναι η Ελλάδα. Και θέλω να σας υπενθυμίσω, στη Βιτεμβέργη το 19ο αιώνα είχαμε την εξής κατάσταση. Στη Βάδη Βιτεμβέργη ήταν τέτοια η πείνα που οι άνθρωποι μετανάστευαν στον μέλλον Δρυνό δρυμό με συγχωρείτε, και ίσως και κάποιοι στην Αμερική. Τόσο κοντά δηλαδή και με τέτοιες διαφορές. Ο Ντάιμλερ παρήματο χάρη, ο Γκότλιπ Ντάιμλερ, και αυτός είναι μια τέτοια περίπτωση που αναγκάστηκε να μεταναστεύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί κανείς να βοηθήσει μια φτωχή επιτροπή να εξελιχθεί οικονομικά, αλλά βέβαια χρειάζεται χρόνος. Και τρίτον, σήμερα δεν είναι τελειωτικό και δεν είναι ε, μη αναστρέψιμο το ότι αυτοί που σήμερα είναι ανεπτυγμένοι ενδεχομένως στο μέλλον να βρίσκονται σε άλλη θέση. Και αυτοί που είναι αδύναμοι θα μπορούσαν να καταστούν οι μηχανή ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι η Ευρώπη και η Νομισματική Ένωση θα βγουν ενισχυμένοι από την κρίση εάν ακολουθήσουμε τα σωστά μέτρα. Με αυτά τα λόγια κλείνω τη σημερινή ε, συνεδρίασή μας και θα μου κάνετε, προσφέρετε χαρά και τιμή αν ε, δεχτείτε την πρόσκλησή μας για τη δεξίωση.